Okay. Um, I'm looking around μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω αν φωνάζει κανείς και να έχει αντίρρηση, οπότε ε, κανένα πρόβλημα. Δεν είμαι και σίγουρη ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Διότι δεν έχουμε τους ε, σκιώδεις ε, για το πρώτο και δεν πρόκειται να κάνω τι ανακοινώσει μου ενώ είναι καινή η αίθουσα. δεν ε, θα αρχίσουμε γιατί δεν έχουμε αρκετούς βουλευτές και αρνούμε σε μια καινή αίθουσα να κάνω εγώ ανακοινώσει και είπαμε ότι για το πρώτο θέμα δεν είναι εδώ οι αρμόδιοι. Ο Ζαμπόλη δεν είναι εδώ. <laughs> δεν έχουμε έλκα εδώ. Άρα δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε. Ε, μα, ε, εντάξει, περιμένω να έρθουν όλες οι ομάδες ε, και οι δικοί σας βεβαίως πάντα. At least one third of our group is represented. Mm. Hm. Μία ομάδα τουλάχιστον είναι εδώ. Μια στιγμή. You're, you're doing S&D, that's okay. Okay, right. Well, in that case... Um, Καλώς. Ε, Περνάμε στο σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών τη 4 Η 5ης η νοεμβριου Υποθέτω πως εγκρίνονται. Θα κάνω τι ανακοινώσει τη Προέδρου όταν ε, έχει έρθει και κάποιο άλλο για να τι ακούσει. Όπω είπα δεν θέλω να μιλάω σε άδεια αίθουσα. Περνάμε σημείο 4 δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία. Η συγγήτρια είμαι εγώ. Και θα εξετάσουμε τις τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα να πω πως υπάρχει σύγκληση με την ε, πλειοψηφία των τροπολογιών, κατά το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε συμβασμούς που θα δεχτεί η πλειοψηφία σκοπεύω να μοιράσω κάποιες πρώτες συμβιβαστικές τροπολογίες μετά από τη λήξη της συνεδρίασης. Επίσης να πω πως υπάρχει τώρα μια γνωμοδότηση, μόνο γνωμοδότηση υπό το άρθρο 49 και όχι το άρθρο 50 γιατί έτσι μαζί με την Γιούρη έτσι προέκυψε αυτό μετά από τις διάφορες μάχες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όριο και είδη δημοσιοποιήσεων. Ε, υπήρχαν τροπολογίες και για να ανέβει και για να κατέβει το όριο. Ε, εδώ πέρα μάλλον τελικά ίσως θα τα η ψηφοφορία τα ζητήματα αυτά. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς το πεδίο εφαρμογής, ειδικά ε, όταν ε, προσπαθούμε να κάνουμε τις εταιρείες να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες ε, από την αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν. Δεν θέλουμε να τις επιβαρύνουμε. Πρέπει να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το βάρος, να βρεθεί μια ισορροπία. Εγώ έλεγα πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε το τζίρο μιας εταιρείας, όχι τον αριθμό υπαλλήλων, ειδικά γιατί οι χρηματοπιστωτικές εταιρείε μπορούν να έχουν μεγάλο τζίρο αλλά αναλογικά λίγους υπαλλήλους, αλλά να έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Οπότε πρέπει, εγώ θεωρώ, να συμπεριλαμβάνεται ο τζίρος, αλλά είμαι διατεθειμένη να δω τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι και να σκεφτούμε την ευθυγράμμιση με την πρόσφατη οδηγία περιλογιστικής. Επίσης άλλες ε, πολιτικές όπως ε, η αλυσίδα εφοδιασμού και η γενική ιδέουσα επιμέλεια πηγαίνει και αυτό προς μια παρόμοια κατεύθυνση για τα διεθνή πλαίσια και πάλι οι τροπολογίες είναι παρόμοιες και κάποιες πηγαίνουν παραπέρα από την αρχική μου πρόταση οι άλλες πηγαίνουν πέρα από την πρόταση να βασιζόμαστε σε κάποιο διεθνές ή ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, κατανοητό, καθώς βεβαίως έτσι βασιζόμαστε σε κατευθυντήρες γραμμές όπως αυτές του ΩΣΑ για τις πολυεθνικές και μάλιστα μια που θα έρθει και ο Γενικός Γραμματέας του ΩΣΑ εδώ πέρα αύριο μπορούμε να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Χαίρομαι που βλέπω πως πολλές τροπολογίες συζητάνε αναφορά αναχώρα, είναι σημαντικό αυτό καθώς σε γενικές γραμμές ε, είμαστε πρωτοπόροι και οπωσδήποτε πιο μπροστά από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να το προωθήσουμε αυτό το θέμα μια που μας στηρίζει η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Και πάλι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Εγώ κατέθεσα κάποιες δικές μου, άλλες ε, τις υπέβαλα αλλού. Υπάρχουν άλλες από τους σοσιαλιστές και οπωσδήποτε είμαι διατεθειμένη να ακούσω και την ε, Αρλίν που ήταν η συγγήτρια στην πρόσφατη οδηγία περί λογιστικής. Ίσως υπάρχει ζήτημα με το να μπει κάπου, μια, κάπου λογικά μια τροπολογία εκεί όπου όντω ανήκει. Ίσως να μην, να μην πρέπει να ανοίξουμε τέτοια ζητήματα Οπότε συμφωνώ πως πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ευρύτερο δυνατό πεδίο εφαρμογή. Οπότε είμαι υπέρ του να, υπάρχει αναφορά, να υπάρχουν αναφορές σαν χώρα και να υπάρχει κάποιος έλεγχος αναφορών. Τώρα, για τις σχετικές απαιτήσει ε, θα πρέπει να τον θαρρύνουν αυτό οι εταιρείε και άρα είμαι υπέρ των σχετικών τροπολογιών μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε σε μια συμβιβαστική πρόταση ή να τις ψηφίσουμε όσο έχουν. Είναι νομίζω σωστό σε αυτή τη φάση η απέτηση αυτή ε, να παραμείνει για τις εισηγμένες ε, εταιρείε. Αλλά και πάλι είμαι ανοιχτή σε προτάσεις. Όσον αφορά τώρα την αρχή συμμόρφωση ή εξήγηση, μου αρέσει αυτή η αρχή για να υπάρχει μια ευελιξία στις εταιρείε, αρκεί να σκέφτονται το τι κάνουν ως προς αυτά τα ζητήματα και το πώς επηρεάζεται η κοινωνία. Πρέπει να δίνουν ξεκάθαρες εξηγήσει, όχι να λένε «Ε, δεν το σκεφτήκαμε, δεν σκεφτήκαμε όταν σημαντικό. Να μην είναι απλά δηλαδή έτσι κάτι το τυπικό. Μετά. Ο Ζαν Πολ Γκοζές... Ε, ε, υπέβαλε μία ρήτρα ασφαλούς ε, λιμένα, καταφυγίου, γιατί εάν εφαρμοστεί λάθος η οδηγία θα μπορούσε να υπάρξει μια ρητρα ασφαλους λιμενα καταφυγείου γιατι αν εφαρμοστει λαθος η εξαίρεση αν ε, υπάρχουν κάποιες αμφισβητήσιμες πρακτικές της δημόσιας διοίκησης όσον αφορά τη διαφάνεια. Βασικό κομμάτι λοιπόν εδώ πέρα βεβαίως είναι ο αντίκτυπο, να πούμε ε, κάτι για τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα. Ειδικά εάν ε, προκύψει γρήγορα και η έκθεση της Κομισιόν. Η προσέγγιση που είχα στην Οδηγία Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 4 είναι να γίνονται οι δημοσιεύσεις, οι δημοσιοποιήσεις και Εάν δεν γίνεται κάπου να δημοσιοποιηθούν στοιχεία, να πάνε τα στοιχεία στην αρμόδια αρχή ή στις αρχές. Αλλά γενικά κατά κανόνα θα πρέπει ε, τα στοιχεία να είναι δημόσια και αν υπάρξει κάποια υπαναχώρηση πρέπει να είναι δικαιολογημένη και ελάχιστη. Νομίζω λοιπόν πως θα είναι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε αυτό και αύριο με τον ΩΣΑ για τις πράξεις κατεξιοδότηση της Κομισιόν για τους ελάχιστους δείκτες. Αναμένω τις δικές σας εξηγήσεις, ε, Φιλίπ, γιατί αναρωτήθηκα γιατί ε, δώσατε στην ε, Κομισιόν περαιτέρω αρμοδιότητες αντί να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις σε ευρωπαϊκό ή διεθνές πλαίσιο. Μετά, υπάρχουν πολλές απορρίψεις της ε, πρότασης από γερμανικές πηγές. Θα μπορούσα να ζητήσω κάποια εξήγηση, αλλά αντιλαμβάνομαι πως η διαφάνεια είναι κάτι που πονάει στη Γερμανία. Επανέρχεται συνεχώς. Συχνά φαίνεται ότι προσπαθούν να την μειώσουν δεν με ενθουσιάζει. Όπως ε, δεν ενθουσιάζει και αυτούς βεβαίως το να κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο ό,τι θέλει στις ε, χρηματοοικονομικές υπηρεσίε. Όλοι λοιπόν πρέπει να συμμορφωθούν εδώ πέρα. Θα περάσω τώρα σκιώδες εισηγητές. Ζαμπολ Γκοζές. Merci Madame la Présidente. Je craignais d'être arrivé en retard, mais je σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σας, το συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα μιλήσω για ένα συγκεκριμένο σημείο για την τροπολογία την οποία έχω υποβάλει και στην οποία αναφερθήκατε. Νομίζω ότι ε, δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε μια τοξική ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι διάβασαν την τροπολογία αυτή. Μάλλον δεν την κατάλαβαν καλά, ενδεχομένως κάποιοι να μην την διάβασαν καν. Υπήρχαν κάποιοι από τις γαλλικές αρχές που ήρθαν και μου είπαν μάλιστα ότι προσπαθώ εγώ να καταρρύψω όλες τις προσπάθειες που προσπαθούμε να καταβάλουμε αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη, δεν ακούω την αγγλική διερμηνία, λέει η Πρόεδρος. Περιμένω λοιπόν να βάλετε τα ακουστικά σας κυρία Πρόεδρε γιατί δεν θα επικοινωνήσουμε διαφορετικά πολύ καλά. Σα έλεγα λοιπόν ότι ορισμένοι μάλλον δεν διάβασαν ή παρανόηση τροπολογία. Διακόπτη πρόεδρο, συγγνώμη, ακούω τη γαλλική διερμηνία στο αγγλικό κανάλι. Μα τι, τι ευτυχία, τι ευτυχία, πραγματικά. Καταπληκτικά, λέει ο κύριο Γκοζέ. Α ε, περιμένουμε. Μια φορά προσπαθώ να έχουμε μαζί σα δημόσιο διάλογο και δεν μα βοηθάει τελικά η τεχνολογία. Ναι, ακούω την αγγλική διερμηνία πλέον, λέει η πρόεδρο. Κύριος Γκοζές, σας έλεγα λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα το εκρηκτικό στο περιεχόμενο της τροπολογίας, με δεχομένως κάποιοι να μην κατάλαβαν καλά τι προσπαθώ εγώ να πετύχω με την τροπολογία αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να στραφώ καθέσον ένα χώρα. Απλώ σε μια συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε κάποιε χώρε όπου οι εθνικέ αρχέ δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών. Υπάρχουν χώρε οι οποίε δεν είναι ιδιαίτερα ανοιχτέ και διδακτικέ και απαγορεύουν τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών. Στην περίπτωση αυτή τι κάνει μια επιχείρηση, τι κάνει μια εταιρεία. Στην τροπολογία μου προτείνω το ακόλουθο αν σε μια χώρα προβλέπεται σχετική απαγόρευση δημοσιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών, τότε η εταιρεία αυτή δεν θα εξαιρείται. Δεν θα προβλέπεται παρέκκληση για την εταιρεία αυτή. Θα πρέπει να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να παρουσιάσει την περίπτωση αυτή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα κρίνει στην περίπτωση, στην συνέχεια, αν αιτιολογείται ε, η παρέκκληση αυτή ή όχι. Η μη δυνατότητα δηλαδή υποβολής ε, πληροφοριών αναδιατυπώνοντας ε, την ε, τροπολογία μου αυτή, θα έλεγα ότι ε, δεν μπορούμε να υποβάλουμε ή να υπάρχει υποχρέωση υποβολής πληροφοριών αν αυτό επισύρει κυρώσεις στη συνέχεια σε ένα κράτος μέλος για μια εταιρεία. Αυτή την περίπτωση ακριβώ προσπαθούσα να περιγράψω στην τροπολογία μου αυτή. Σε καμία περίπτωση θέλω να δημιουργήσω μια περαιτέρω εξαίρεση. Λέω απλώ ότι για τι χώρε εκείνε όπου προβλέπεται απαγόρευση δημοσιοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών από τι εταιρείε, θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη που θα κρίνει τι θα πρέπει να συμβεί με τι εταιρείε αυτέ. Αυτά είχα να σα πω. Σα έχω κατά τα άλλα απόλυτη εμπιστοσύνη, κυρία Πρόεδρε. Okay, thank you very much. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. μιλώ ονόματο τη της ε, ομάδας μου. Έχω και προσωπικέ παρατηρήσει, αλλά αρχίζοντα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, νομίζω είναι πολύ καλή η γνωμοδότηση. Ευχαριστώ και με όλου του προλαλήσαντε. Είναι σημαντικό η Επιτροπή μα με ξεκάθαρο τρόπο να ορίσει τι θα θέλαμε να προβλέπετε για την δημοσιοποίηση, πέρα από αυτά που έχουμε κάνει ήδη για την ε, κοινωνική, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχουμε βασικούς ε, δείκτες ε, επιδόσεων, ε, έχουμε ισχυρή αρχή του, της συμμόρφωσης ή εξήγησης, αιτιολόγηση, όπως μας είπε και ο εισηγητής. Χαιρόμαστε για, τα περί διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού. Μας ικανοποιεί μεγαλύτερη διαφάνεια για τις φορολογικές ρυθμίσεις. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα αμφιλεγόμενα, σοβαρά αμφιλεγόμενα ζητήματα, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συνένεση και θα καταθέσουμε μια ισχυρή έκθεση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, όπου είμαι επίσης μέλος, ε, με τον Κλάους, λένε ε, είχαμε ασχοληθεί με την οδηγία διαφάνειας ε, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και τώρα θα ήθελα να στραφώ στο Ζαν Πολ. Δεν θα ήθελα να εξετάσουμε το ζήτημα των ποινικών κυρώσεων για όλους τους τομείς της βιομηχανίας. Το πρόβλημα που έχω είναι αν ξανανοίξουμε τα συμπεφωνημένα, δηλαδή αυτά που ισχύουν για τη δασοκομεία και την εξωτερική βιομηχανία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί έχουμε παγκόσμιους ε, κανόνες. Έχουμε την νομοθεσία του Frank στη ΣΥΠΑ. Δεν μπορούμε τώρα να ξανοίξουμε αυτά τα κεφάλαια, όχι μόνο ε, διότι υπογράψαμε αυτή την νομοθεσία όταν ήρθε η Άγξουσή για να παραλάβει το βραβείο Ζαχάροφ και τότε είπε σε συνεντεύξει τέλο πάντων που έδωσε, είπε ότι ε, στη Βυρμανία έχουμε πλούσιου πλουτοπαραγωγικού ε, πόρου, ε, πετρέλαιο και το καθεξής. Οπότε για τις αναπτυσσόμενες χώρες τα περί εξορρεκτική βιομηχανία έχουν μεγάλη σημασία και Ζαν Πολ το τονίζω, δεν μπορούμε να ξανανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο της ε, γιατί απερίφθη δικαίως από τις ΗΠΑ διότι εάν να ε, ε, ε, επιτρέψουμε τέτοιες αποκλήσεις, το Καμερούν, η Αγγόλα και άλλες τέτοιες χώρες θα μπουν στο παιχνίδι και δεν θα επικρατεί πλέον διαφάνεια. Δηλαδή θα ρίξετε μια τεράστια τρύπα στο νέο σύστημα. Ήταν ατελείωτες ε, οι διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο και οι μεγάλες ε, πετρελαϊκές εταιρείες ε, έχουν στείλει μία επιστολή που δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση. Θελημένα, εσκεμμένα αυτές οι εταιρείες δεν θέλουν ε, να καλυφθούν οι υπόλοιποι τομεί. Θέλουν να ξανανοίξει το κεφάλαιο τη εξορρυκτική βιομηχανία γιατί είναι προ ε, συμφέρον του. Πρέπει να το αποφύγουμε αυτό πάση θυσία ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ατυχώ μα καλεί να υιοθετήσουμε την ίδια προσέγγιση για όλου του τομεί. Τέλο πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο εισηγητή κάνει μια καλή, προτείνει μια καλή ενδιάμεση λύση μέσα σε συγκεκριμένο άρθρο να προτείνουμε τι εκθέσει ανα χώρα για όλους τους βιομηχανικούς τομέας, αλλά το φυσικό αέριο, τον, το πετρέλαιο και την εξωτερική βιομηχανία ας τα αφήσουμε στην άκρη, διότι είναι πολύ διαφορετικός αυτός ε, ο τομέας και ξαναλέω ε, στις αναπτυσσόμενες χώρες θα κάνουμε, θα ανοίξουμε το παράθυρο για όλα τα διεφθαρμένα καθεστώτα για να μην δημοσιοποιούν καμία πληροφορία. Όχι, ε, πρέπει να ισχύουν διαφορετικά πρότυπα για αυτό το κλάδο. Τώρα, προσοχή, κρούτων, κόδωνα του κινδύνου όχι επειδή θέλουν να δημιουργήσω δυσκολίες, αλλά επειδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι δύσκολο το ζήτημα, τελειώνει η θητεία μας ε, και στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου θα έχουμε τρεις προτάσεις. Η μία δεν θα αναφέρεται καθόλου στο CSR, e ε, αυτό, αυτή ε, το Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα έχουμε την πρόταση της Προεδρίας που μου αρέσει εν μέρη, είναι ισχυρή, υπάρχει έλεγχος και μέσα στην οικονομική δήλωση θα έχουμε και μη χρηματοοικονομική σε πληροφορίες, οπότε θα έχουμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Μπορούμε βεβαίως να ε, την κάνουμε πιο ήπια την πρόταση, αλλά θα είναι υψηλό το αρχικό πρότυπο και η τρίτη πρόταση θα είναι η πρόταση του εισηγητή και του Μπαλτασέρη, που είναι αποδυναμωμένη, είναι ασθενέστερη ως προς την νομοθετική κατοχήρωση και κάποιοι θα πούνε ότι αυτό που δεν θέλουν είναι όλες οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες να αποκλειστούν γιατί δεν μπορούμε εμείς να συμφωνήσουμε για τις ε, εκθέσεις αναχώρα, το CBSCR. E ε, και ε, Όντω είναι μεγάλο το διακύβευμα σε αυτό το τομέα, αλλά ο εισηγητή με του σκιώδει θα πρέπει να ε, σκέφτονται στρατηγικά με ποιο τρόπο θα έχουμε την καλύτερη προσέγγιση για να επιτύχουμε την καλύτερη συμφωνία και αυτό που ε, δεν πρέπει να επιτρέψουμε είναι να υπονομεύσουν κάποιες ε, βιομηχανίες ε, το όλο εγχείρημα για να ξεφορτωθούν εντελώς τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης και υποβολής αναφορών αναχώρα. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Η Επιτροπή μας, ο εισηγητής και κατά επέκταση η Επιτροπή πρέπει να καταθέσει μια ισχυρή πρόταση. Πολλοί νιώθουν ιδιαίτερο σκεπτικισμό και δεν θέλουν να περάσουν όλες αυτές οι προτέσεις και σίγουρα δεν πρέπει να κάνουν το παζάρι με του συναδέλφου, ε, να του δώσουν τι εκθέσει αναχώρα για να δώσουν οι υπόλοιποι τις μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Όχι, δεν πρέπει να γίνει αυτό το παζάρι. Ε, Πρόεδρος, ευχαριστούμε και ε, χαιρόμαστε μπορούμε να υποφεληθούμε από την εμπειρία σα, Φίλιπ. Uh, uh, σε σχέση με αυτά που είπε η Ερλίν, καταρχά, πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να προστατεύσουμε τη δυνατότητα υποβολή εκθέσεων αναχώρα και να συμπεριλάβουμε τόσο την εξορρυκτική βιομηχανία αλλά και τις τράπεζες. Ξέρετε ότι το ζήτημα αυτό πρέπει εμείς να το προωθήσουμε, να μην το αφήσουμε αποκλειστικά στο G20 και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εξαφανιστεί από την πρόταση. Και συμφωνώ επίσης με τα υπόλοιπα τα οποία πρότεινε η Αρλίνα. Το να δώσουμε κάποιες ειδικέ εξαιρέσεις θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλές χώρες όπως είπε, στην Αγκόλα αλλά ακόμα και στα νησιά Κέιμαν να επωφεληθούν από την εξαίρεση αυτή και να μην τελικά γίνει απαραίτητη δικαστική έρευνα που θα έπρεπε να γίνει, καθώς επίσης και η επιβολή κυρώσεων για τις χώρες αυτές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει η υποχρέωση αυτή να προβλέπεται για όλους, η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων να χώρα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προβλεφθούν και υψηλότερε κυρώσεις από τις δικαιοδοσίες δοσίες εκείνες με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Τουλάχιστον υπάρχει μία εναρμονισμένη προσέγγιση προς αυτό και να δώσουμε κατά αυτόν τον τρόπο τα απαραίτητα κίνητρα στις επιχειρήσεις για να λειτουργούν σωστά. Όσον αφορά τώρα τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Όταν διαπραγματευόμασταν την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων, νομίζω ότι περισσότερες χώρες ήταν κατά της δικής μας προσέγγισης, με την εξαίρεση ενδεχομένως της Γερμανίας, αν θυμάμαι καλά. Ουδής ήταν πάντως υπέρ μας. Πλησιάζουν πάντως οι ευρωπαϊκές εκλογές και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη στάση που κρατάμε απέναντι στην κοινή γνώμη. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ε, πώς μπορεί ποτέ οποιαδήποτε κυβέρνηση να δικαιολογήσει μια στάση κατά της διαφάνειας. Ξέρετε ότι υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα υψηλότερο επίπεδο γραφειοκρατίας. Ξέρετε ότι δεν ισχύει όμως κάτι τέτοιο. Ξέρετε ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τα αριθμητικά αυτά δεδομένα, τα έχουν στη διάθεσή τους δεν ε, χρειάζεται να καταβάλουν καμία απολύτως προσπάθεια προκειμένου να δημοσιοποιήσουν τα δεδομένα αυτά. Επομένως δεν μπορώ να αποδεχθώ καμία απολύτως δικαιολογία από κανέναν Υπουργό Οικονομικών ο οποίος θα ταχθεί κατά της δημοσιοποίησης των δεδομένων αυτών. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε και το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια του οποίου το Συμβούλιο θα πρέπει να τηρήσει την υπόσχεση την οποία έδωσε το Μάιο όταν είπε ότι μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι αυτό το Δεκέμβριο του 2013 θα είχαν καταργήσει εντελώ το τραπεζικό απόρριτο. Εμεί μπορούμε πλέον να ασκήσουμε περισσότερη πίεση και να πούμε προ υπουργού πραγματικά θα διατηρήσετε την υπόσχεσή σα όσον αφορά το τραπεζικό απόρριτο και αν τελικά εφαρμόσετε όντω την υπόσχεσή σα αυτή, θα ταχθείτε κατά τη υποβολή εκθέσεων χώρα και πραγματικά επιθυμείτε ένα δημόσιο διάλογο για το ζήτημα αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί έτσι ώστε ναι μεν να μην στραφούμε κατά της δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, αλλά και παράλληλα να στείλουμε το σωστό μήνυμα προς την κοινή γνώμη. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ορισμένοι προσπαθούν πραγματικά να δικαιολογήσουν πράγματα καθαρά δικαιολόγητα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει και εμείς να διατηρήσουμε μια στάση πολύ πιο ισχυρή. Ξέρουμε ότι στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε πολύ καλούς συναδέλφους οι οποίοι μπορούν να ασκήσουν επιρροή και ξέρετε ότι με την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων δεν χρειάστηκε να λάβουμε υπόψη μας τη γνωμοδότηση της ε, Γιούρη. Αυτή τη φορά βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Θα έλεγα πάντως και προς συναδέλφους ε, της Γιούρη το ίδιο πράγμα. Ο κύριος Λένε πραγματικά θέλει να εμφανιστεί ως ε, υπερασπιστής της αδιαφάνειας. Σαφώς μπορεί να πει κανείς ότι έχουν περάσει πια οι γερμανικές εκλογές, αλλά και πάλι αυτό δεν θα δικαιολογούσε μια τέτοια στάση. Εγώ είμαι πάντως έτοιμος να εκθέσω τους συναδέλφους αυτούς και να διατηρήσω μια πολύ ισχυρή στάση. Τώρα, πώς μπορεί να γίνει πιο αποδεκτή η πρόταση αυτή. Ορισμένοι λένε ότι η εφαρμογή της υποβολής εκθέσεων χώρα και όλων των υπόλοιπων διατάξεων για τις μικρές επιχειρήσεις αυτό όντως μπορεί να προκαλέσει ένα περαιτέρω άκθος. Εμείς προτείνουμε μία σταδιακή προσέγγιση σε τρία βήματα, σε τρία στάδια. Προβλέπουμε δηλαδή τρία επίπεδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα επίπεδο κάτω του οποίου α, εξαιρείται κανείς από τις υποχρεώσεις της νομοθεσίας. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρώτο στάδιο το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί στο μέλλον. Πάντως για τις πιο μικρές επιχειρήσεις θα προβλέπεται μία εξαίρεση. Στο δεύτερο στάδιο θα ισχύει το συμμόρφωση εξήγηση και στο τρίτο επίπεδο η συμμόρφωση θα είναι πλέον υποχρεωτική. Και πιστεύω ότι εμείς μπορούμε να καταφέρουμε να βρούμε τον κατάλληλο συνδυασμό όλων αυτών των τριών επιπέδων συμμόρφωσης που σας εξήγησα και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τα σωστά όρια. Και αυτό θα αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα προκειμένου να γίνει αποδεκτή δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τους περισσότερους συναδέλφους. Τώρα, όσον αφορά τις κατεξοδότηση πράξης Σάρων, θα μπορούσε να μου δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ποιο σημείο ακριβώ δεν ε, συμφωνήσει. Εγώ ουσιαστικά έλεγα ότι θα έπρεπε να είχαμε κοινά πρότυπα δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Εσύ πιστεύει ότι τα πρότυπα αυτά πρέπει να μπουν στο διατακτικό και να μην προβλέπονται απλώ στι ε, κατεξτότητε πράξη, Πρόεδρο. Θα το σχολιάσω αυτό λίγο αργότερα. Η ερώτησή μου είναι η ακόλουθη. Πώς μπορεί να συνδυαστεί η πρότασή σου αυτή με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσουν είναι γενικότερο κάπως το πρόβλημα. Άσλι. Ε, um, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα μου σε γενικές γραμμές υποστηρίζει την αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν. τώρα ακούω Ιταλικά. Ε, buongiorno, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, λειτουργεί. Ακούτε αγγλικά. Λοιπόν, ωραία. Να ξεκινήσω πάλι. Η ομάδα μου σε γενικές γραμμές υποστηρίζει την αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν και την προσέγγιση, συμμόρφωση ή εξήγηση. Αυτό το οποίο δεν υποστηρίζουμε είναι πολλές τροπολογίες που κυρίως προέρχονται από τα αριστερά της εύσας οι οποίες απλά προσθέτουν ε, αχρίαστες ε, ρυθμίσεις. Να υπενθυμίσω στον κύριο Λαμπέρ ότι οι εταιρείε αυτές που περιγράφει ως σατανικές ε, απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους, έχουν κέρδη, τα κέρδη φορολογούνται, οι φόροι πληρώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες και τα, τα μερίσματα πάνε στους συνταξιούχους μας. Μα εγώ θέλω να λειτουργήσει σωστά το σύστημα, λέει ο κύριος Λαμπέζ. Ωραία. Κοιτάξτε. Οι μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν στόχο να συμπληρώσουν πράγματι τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Σωστό αυτό για τις εισηγμένες, αλλά για ιδιωτικές εταιρείες δεν ξέρω τι χρειάζεται, καθώς δεν έχουν τον ίδιο αριθμό επενδυτών. Βεβαίω, ε, οτιδήποτε θέλουν οι επενδυτές τους μπορούν εθελοντικά να το δώσουν αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθούν οι προτάσει αυτές σε μικρομεσαίες επιχειρήσει. Όσον αφορά την ε, πολυμορφία Βεβαίω αναγνωρίζω μια σχέση μεταξύ της ανθεκτικότητας μιας εταιρεία και της πολυμορφίας του ΔΣ. Αλλά αυτό θα το άφηνα εγώ στι ίδιε εταιρείε παρά στη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών. Συμφωνώ όμως με τον συνάδελφο του ΕΛΚ Σαριουσέα, πως εδώ πέρα έχουμε κάποια πράγματα που αλληλεπικαλύπτονται με την οδηγία περί ισότητας και παραβλέπουμε τα εθνικά πλαίσια που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Επίσης, ε, είμαι κατά άλλων διακρίσεων πέρα του φύλου που ήδη αναγνωρίζονται στο ευρωπαϊκό δίκαιο, όπως παραδείγματο χάρη γεωγραφική πολυμορφία, μορφωτική πολυμορφία και, ε, ε, και επαγγελματική εμπειρία. Όλα αυτά είναι μπουρδες κατά την άποψή μου. Όσον αφορά δε τις αναφορές αναχώρα, όσον αφορά την φορολογία, δεν θεωρώ πως χρειάζονται καθώς είναι δυσερμήνευτες αυτές οι απαιτήσει και θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Βλέπω πως το κομμάτι αυτό δεν το συνοδεύει κάποια αξιολόγηση αντικτύπου. Κυρία Πρόεδρε, θα τελειώσω εδώ. Απλά θα πω πως ελπίζω οι προτάσεις της Κομισιόν να μην ξεχυλώσουν προς τα αριστερά από την Επιτροπή μας. Το αποτέλεσμα θα είναι λιγότερες δουλειές, λιγότερη ευημερία και περισσότερες θέσεις εργασίας που θα πάνε εκτός Ένωσης. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Κάποιος άλλος. Βόλφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποια σχόλια. Φίλιπ, ε, εμείς πρέπει να κάνουμε το σωστό, όχι αυτό το οποίο θέλει, θέλει κοινή γνώμη. Ναι, ναι, καμιά φορά συμπίπτει, ναι. Πάλι γαλλικά ακούω, λέει η πρόεδρος. Κάτι, κάτι φυτό φρικτό συμβαίνει με τα κουμπιά στην αγγλική καμπίνα, δεν ξέρω. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μιλήσετε λίγο. Ωραία, λοιπόν. Κάποιες γερμανικές εταιρείε στο παρελθόν στο μηχανολογικό τομέα πράγματι δεν συμπεριφέρθηκαν σωστά και αυτό βεβαίως είχε ως αιτία τη γερμανική φορολογική νομοθεσία που επέτρεπε στις εταιρείε να θεωρήσουν τις μίζες ως πληρωμές δημοσίων σχέσεων. Ναι, ναι, έτσι, έτσι ήταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Και Βεβαίω, όταν έχουν μάθει έτσι, αυτό δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη, ανεξαρτήτως του τι οδηγίε θα περάσουμε. Οπότε, αντί τώρα να αλλάξουμε ολόκληρο τον κλάδο και τις μικρομισές επιχειρήσεις, εγώ θα επικεντρωνόμουν στο κομμάτι που πιθανότατα ακόμα κάνει ζαβολιές, πέρα από τις εξορρυκτικές κλπ ε, το τα μηχανολογικά έργα. Εκεί πέρα όταν υπάρχουν μεγάλα έργα, φτιάχνει κανείς εργοστάσια, ε, η πιθανότητα για μίζες ε, είναι υψηλή. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Συμφωνώ με όλους τους στόχους, αλλά ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα και το αποτέλεσμα δεν θα είναι ικανοποιητικό. Οπότε... Εγώ θα προσέθετα και τον τομέα των μηχανολογικών και των μεγάλων δημοσίων έργων και τέλος. Ε. Μάλιστα. Όλε Λούτβιξον, ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρόταση νομοθετήματο κατά τη γνώμη μου. Πολλέ μεγάλε επιχειρήσει ε, φέρουν μεγάλη ευθύνη και πρέπει να την επομιστούν και για το περιβάλλον αλλά και για τα κοινωνικά ζητήματα και την ποικιλομορφία. Ε, το νομοθετικό πλαίσιο είναι και το λογικότερο πλαίσιο, αν θέλετε, για να ρυθμίσουμε τη διαδικασία. Τέσσερις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Πρώτα απ' όλα, ε, θα πρέπει ε, να καλυφθούν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, από ένα συγκεκριμένο κύκλο εργασίας και πάνω και από ένα συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων και πάνω. Στη συνέχεια για την επικοινομορφία είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει τέτοια η δημοσιοποίηση. Τρίτον, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται οι πληροφορίες για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, ακόμη και αυτά που συμβαίνουν σε επίπεδο υπεργολάβων. Τέταρτον, οι εταιρείε θα πρέπει να ενημερώνονται ε, για οποιαδήποτε απόκληση ε, ως προς τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία σε οποιοδήποτε σημείο της αλυσίδας. Στη συνέχεια για τις εκθέσεις αναχώρα και το προτινόμενο σύστημα σε εκθέσεων θα πρέπει να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις σε όλους ε, τους τομείς. Ε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οποιαδήποτε είδους εξαιρέσεις. Θα πρέπει ε, λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τον κοινό νου για να καταλήξουμε σε ένα λογικό κείμενο που θα γίνει αποδεκτό από όλους. Right, now Ευχαριστώ. Ο Φιλίπ μιλάει στο τηλέφωνο, αλλά σε πιάσα τα πράσα, αλλά θέλεις να μιλήσεις. Ε, Πολύ μ' αρέσει ο πολιτικός διάλογος, αλλά δεν μ' αρέσει να ακούγονται ψευδή πράγματα. Εγώ δεν είπα ε, να ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις για όλους, ακόμη και για τις ΜΜΕ. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι τριών ταχυτήτων το σύστημα και θυμάστε τι είχα πει για τις μικρομεσαίες. Όταν συζητούσαμε τις λογιστικές οδηγίες και την οδηγία για τη διαφάνεια, είπαμε ότι πρέπει να ισχύσει το διπλάσιο όριο σε σχέση με τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπάρχει ένα όριο κάτω του οποίου δεν ε, χρειάζεται δημοσιοποίηση περισσότερων πληροφοριών. Θα υπάρχει αυτό το πρώτο στάδιο. Δεύτερον, όπως είπε και ο Βόλφ, ε, μιλάμε ναι, όντως για τη διαφθορά. Όμως, όταν μιλάμε για την υποβολή εκθέσεων αναχώρα και μιλάμε για τις έξι βασικούς δείκτες ε, που έχουμε ήδη επιβάλει σε άλλους τομείς, αυτό επιδιώκουμε διαφάνεια και για τα φορολογικά ζητήματα. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο θα ήταν δύσκολο. Εγώ ε, στην IBM δούλευα και εκεί είχαμε στοιχεία ε, ανά χώρα. Δεν ε, απαιτείται καμία προσπάθεια, μηδενική προσπάθεια απαιτείται για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών. Εντάξει, άλλο το αν θα το δεχτούν οι εταιρείε, αλλά δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Ούτε παραπάνω λογιστέ, ούτε παραπάνω μεγαλύτερο οικονομικό έλεγχο, μόνο δημοσιοποίηση χρειάζεται. Συγγνώμη, Άσλη, αν πιστεύει ότι αυτό απειλεί τον καπιταλισμό τότε θα καταλήξω στο συμπέρασμα. Συγγνώμη, ε, ο Άσλη εκτό μικροφώνου λέει ότι δεν είναι δική σου δουλειά. Ε, σοβαρά, δεν είναι δική μου δουλειά να ξέρω πού πληρώνουν φόρους οι εταιρείε. Ε, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ε, δηλαδή η κερδοφορία των εταιριών δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, δεν, δεν, πρέπει, δεν δικαιούμαστε εμείς να γνωρίζουμε πού πληρώνουν φόρους. Μ, μάλιστα. Πολύ ωραία, γιατί δηλαδή ε, βάσει της δικής σου φιλοσοφίας ε, και οι συντηρητικοί πάντοτε υπεραμείνονται της δημοκρατίας και συνήθως σας ακολουθώ κιόλας ε, σε αυτά που λέτε, αλλά sorry, όταν δεν μπορούμε να είμαστε υπεράνω της δημοκρατίας, έχουμε δηλαδή, τι, οι εταιρείε θα συμμορφώνονται με τις κανόνες που θα θεσπίζουν οι ίδιες. Έχουμε δηλαδή τη, τη, τους κανόνες των εταιριών ε, και τι, η δημοκρατία πρέπει να είναι υπόλογης εταιρεία και όχι το αντίστροφο. Ε, συγγνώμη, αλλά ε, μπορεί, Ε, τέλος πάντων διαφάνει για, τους, ε, για τις βασικές ε, παραμετρούς, δηλαδή πόσοι, πόσους που, σε ποιες χώρες δραστηριοποιείται, ποιες είναι οι νομικές οντότητες, ιδιωτικές εταιρείες ή συγμένες εταιρείες, ποια είναι η κερδοφορία σας, όλα αυτά είναι υπό της δημοκρατίας. Υπάρχει μια απέτηση διαφάνειας και δικαίωμα διαφάνειας. Τι, αν έχετε πρόβλημα, σας παραπέμπω και στον Άνταμ Σμιθ. Οι βασικοί παίκτες της αγοράς πρέπει να τα ξέρουν αυτά. Και δεν πρέπει να υπάρχει ασυμμετρία σε σχέση με την ε, χορήγηση πληροφοριών. Όλοι θα πρέπει να ξέρουν τα πάντα για όλους. Ε, και είμαι κι εγώ πολίτης ε, και μπορεί να επιλέξω εγώ να συναλλάσσομαι με εταιρείε που έχουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και όχι με οποιονδήποτε. Αυτή είναι η διαφωνία στην αγορά. Και αν οι εταιρείε δεν μπορούν να δεχθούν το ότι οι πελάτες τους θέλουν να ξέρουν τι κάνουν, δεν πρέπει να είναι στην αγορά, δεν πρέπει να είναι. Ε, εταιρείε. Ή θα πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και θα πιστεύουν ότι είναι καλό και για το γενικό καλό ή αλλιώ πρέπει να αποσυρθούν. Δεν, δεν μπορούν δηλαδή να καταργήσουν την δημοκρατία από την ε, κοινωνία. Δεν μπορούμε δεν, να, δεν μπορούμε να μην, να ξέρουμε πώς παίρνουν μια πρόσοδο από την ίδια την κοινωνία αυτές οι εταιρείε. Άλλος. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ. Ελπίζω να ε, μπορέσω να καταθέσω συμβαστικές ε, τροπολογίες ε, οι οποίες θα είναι ουσιαστικές αλλά όχι και υπερβολικές διότι αυτή είναι η λεπτή γραμμή για να ε, προχωρήσουμε όχι να είμαστε υπερβολικά μαλθακοί αλλά να υπάρχει μια αναλογικότητα να τηρείται αυτή η αρχή νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όπως είπε και η Αρλίν κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να γίνει και δημόσια σύντηση στα κράτη-μέλη στα ΜΜΕ διότι ε, δεν, το θέμα της φορολογίας δεν είναι μόνο ζήτημα πλέον ε, των αναπτυσσομένων χώρων. Εντάξει, θα καταλαβαίνω αυτό που λέτε για την υλοτομία και την εξορρυκτική, αλλά τώρα πλέον πλήττει αυτό το ζήτημα και τις ανεπτυγμένες χώρες. Οπότε πολλές χώρες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε πρόγραμμα λιτότητας ε, και δεν μπορούν να εισπράξουν τους φόρους που δικαιούνται. Για την επιθετική τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και άλλα τέτοια συναφή ζητήματα είναι σημεία που μας βοηθούν διότι είναι συνενετικά. Όμως δεν επαρκούν. Ε, δεν επαρκούν για να γνωρίζουμε πού ε, πρέπει να ξεκινήσει μια έρευνα για ποια εταιρεία, σε ποιο τομέα. Άρα δεν πρέπει να υποχωρήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Καταλαβαίνω δε γιατί ε, έκανε αυτή την πρόταση ο Ζανπόλ και ενστικτοδός κάποιος ε, πιστεύει ότι πρέπει να αποσυρθεί αυτή τη διάταξη γιατί δεν πρέπει κάποιος αδίκος να, ε, ε, να απαγγελθεί μάλλον μια κατηγορία ποινικού δικαίου σε κάποιον αδίκος. Όμως κάποιες χώρες δεν μπορούν να προστατεύονται εφαρμόζοντας μια κακή νομοθεσία και παρεμποδίζοντας τη διαφάνεια. Και το άλλο είναι ότι χρειαζόμαστε τη διαφάνεια και πρέπει να ε, θεσπίσουμε τις κατάλληλες διατάξεις, αλλά ε, οι εταιρείε που θέλουν ε, συμβόλαια Συμβάσει σε αυτές τις χώρε πρέπει να το δεχτούν ότι θα πρέπει να είναι πιο διαφανή. Ε, και στην Ευρώπη ε, θα ε, επεκταθεί αυτό το φαινόμενο ότι είμαστε εμεί η μεγάλη αγορά και περιμένουμε να κάνουν οι άλλοι γενναίε κινήσει για τι διεθνεί συμφωνίε. Περιμέναμε ήδη και ντροπή μα στην Αμερική να βγάλει το φίδι από την τρύπα για την εξορρυκτική. Λοιπόν το έκαναν εκείνοι, Α η σειρά μα είναι να κάνουμε κι εμεί το βήμα που πρέπει να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω ε, οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων να δείξουν και λίγη περισσότερη πυγμή. Αυτά. Ε, τα, το πρώτο σχέδιο θα σας έρθει σύντομα. Αλλά έχω μια σειρά τιμερών διαλόγων και δεν ξέρω πότε θα έχω καιρό για να τα πούμε κάτι ιδιαίτερα, αλλά θα κυκλοφορούν διάφορα έγγραφα για να ξέρουμε οι μεν τι λένε οι και ελπίζω ε, να, να τα καταφέρουμε. 9 Δεκεμβρίου θα ψηφίσουμε. Ε, θα δούμε τι κάνει και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ε, της οικονομίας. Καλά δεν τα λέω, ε. Ο Βόλφ, ε, κλείνει συνεργασίγητης. Ευχαριστώ. Ψάρων, ελπίζω να μ' ακούς. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, χαιρετίζω πρώτα απ' όλα την πρωτοβολία της Κομισιόν να ξεκινήσει μια ευρύτατη συζήτηση για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να έχουμε τα επόμενα χρόνια κάποια πρόβλεψη για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ευρωπαϊκής οικονομίας, γιατί οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις ε, δημιουργούν θέσει εργασίας ε, και διατηρούν την ανταγωνιστικότητα. Εκεί πέρα λοιπόν είναι πίσω αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Θα θυμάστε όλη τη στρατηγική της Λισαβόνας, που είχε ως στόχο το 2010 να γίνει η πιο ανταγωνιστική οικονομία του κόσμου η Ευρώπη. Οπότε δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή εξαρτάται πάρα πολύ από τη χρηματοδότηση των τραπεζών. Ε, κατά 70% σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου είναι αντίστροφη η αναλογια ειναι Ένα 25-30% είναι χρηματοδότηση τραπεζική των επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Δεν ναι, θα μπορέσουμε βέβαια να τα αλλάξουμε εντελώ και δεν θέλουμε κιόλα, αλλά πρέπει παρόλα αυτά να αναγνωρίσουμε πω η βάση μακροπρόθεσμη ε, χρηματοδότηση πρέπει να διευρυνθεί. Όταν πάει κανεί εκτό Ευρώπη και ρωτάει να του πούν την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούει συνέχεια «Ε, είστε πλούσιοι ε, γυράσκεται και άρα αποφεύγεται τον κίνδυνο. Δεν είναι ιδεώδης η κατάσταση. Πρέπει να επενδύσουμε σε εκπαίδευση, τεχνολογία, έρευνα και ανάπτυξη, συγκοινωνίες, τηλεπικοινωνίες για να σταματήσει ε, θα έλεγα η ε, παρακμή και να παραμείνουμε στην πρωτοπορία. Βεβαίως δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από τις παραδοσιακές εμπορικές τράπεζες να κάνουν κάτι τέτοιο, ούτε και από τους χρηματαγορές. Πρέπει εδώ πέρα να συμπράξουν όλοι. Οι ε, επιχειρηματικές τράπεζες, είτε είναι τα ταμιευτήρια, είτε ιδιωτικές τράπεζες, είτε οτιδήποτε άλλο, θα εξακολουθήσουν βεβαίως να είναι ο σημαντικότερος τομέας ε, χρηματοδότησης. Μετά έχουμε τις λεγόμενες αναπτυξιακές τράπεζες. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν αρκετά μεγάλες τέτοιες, όπως η KfW στη Γερμανία, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδόμησης και Ανάπτυξης μπορούν βεβαίως να βοηθήσουν έτσι ώστε μαζί με τους ιδιώτες επενδυτές να έχουμε κάποια μακροπρόθεσμα έργα. Θεωρώ εδώ πέρα πως πρέπει στο πλαίσιο των βέλτιστων πρακτικών ε, κάποιες χώρες ε, να εμβαθύνουν ε, στις εφιστάμενες πρακτικές, να υπάρξουν κάποιες αναπτυξιακές τράπεζες. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει τώρα μια πράσινη επενδυτική τράπεζα, στην Ανταλουσία υπάρχει μια αναπτυξιακή τράπεζα, στην Ιταλία σε άλλη μια χώρα υπάρχουν κάποιες προσεγγίσεις μαζί με την ΚΑΕΦΒ ε, για να ιδρυθούν ε, τέτοια ιδρύματα που θα εργάζονται όπως η ΚΑΦΕ. Οι θεσμικοί επενδυτές, ε, που, στους οποίους παραδοσιακά στρεφόμασταν, είναι σε δύσκολη θέση. Αν σκεφτούμε τις ασφαλιστικές εταιρείε μέσω των ρυθμιστικών απαιτήσεων, δηλαδή της δεύτερης οδηγίας περί φερεγγιότητας ε, έχουν μεγάλες δυσκολίες. Εδώ πέρα λοιπόν η Κομισιόν προσπαθεί μέσω του ΕΛΤΗ να δημιουργήσει ένα ταμείο μακροπρόσωπων επενδύσεων από θεσμικούς επενδυτές επιπλέον. Θα πρέπει να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις ε, να ε, βρουν χρήματα στην αγορά και υπάρχουν βεβαίως και άλλες προσεγγίσεις. Υπάρχει ένα κομμάτι που κάνει ειδικά ε, εισαγωγές στο χρηματιστήριο για μεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, θα πρέπει να προσελκύσουμε και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και ιδιωτικά κεφάλαια και βλέπω στη χώρα μου πως και μεσαίες επιχειρήσεις ε, εκδίδουν δικά τους ε, χρεόγραφα. Και με αυτόν τον τρόπο αυτό το οποίο χρηματοδοτούσαν οι ίδιες οι τράπεζες ε, ε, το κάνουν οι επιχειρήσεις οι ίδιες. Βεβαίως οι τράπεζες προσπαθούν να ισοσκελίσουν αυτή τη στιγμή τους ισολογισμούς τους ε, και βρίσκονται σε μια φάση απομόχλευσης. Επίσης, πρέπει να προσελκύσουμε και τους μικρούς επενδυτές, γιατί εξακολουθούμε σε πάρα πολλές χώρες να έχουμε ε, μεγάλες αποταμιεύσεις. Και με τις δυνατότητες που έχουν οι μικροαποταμιευτές ε, δεν είναι ικανοποιημένοι, γιατί αν πάνε τα λεφτά τους στην τράπεζα έχουν ελάχιστες στόχους και πάρα πολλοί πράγματι φοβούνται να μπουν στις μετοχές ε, ή στα ταμεία, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό ταμείο για μικροεπενδυτές που θα εκμεταλλεύεται αυτή την υφιστάμενη ρευστότητα και θα τη διοχετεύει βεβαίως ε, στις επιχειρήσεις αλλά βεβαίως αυτό θα γίνει με την δυνατότητα μέσω πρόθεσμα κάποιος να αποδεσμευτεί από αυτή του την τοποθέτηση. Ένα θέμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι το θέμα της ε, τιτλοποίησης, ε, το οποίο βεβαίως ε, ε, προκάλεσε μεγάλες ζημιές και μέσω της φούσκας των ακινήτων στην Αμερική, αλλά η τιτλοποίηση από μόνη της δεν είναι κάτι θετικό ή αρνητικό. Αν δεν οδηγεί από τιτλοποίηση σε τιτλοποίηση του ίδιου πράγματος, αν πρόκειται για κάτι το οποίο γίνεται μία φορά, νομίζω μπορεί να είναι κάτι το πολύ λογικό και πρέπει να ενθαρρύνουμε την ε, Κομισιόν να δει το τι κάνει η Γιώσκο και το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής ε, Σταθερότητας. Και βεβαίως υπάρχουν και τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία τα οποία μπορούν ε, κάλλιστα να προσφέρουν δυνατότητες χρηματοδότησης. Συνολικά βεβαίως ισχύει το εξής. Όταν μιλάμε για μακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις, θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε αυτό το κεφάλαιο ειδικά όταν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν έχουμε ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις. Αυτό το σχετίζεται μόνο με τις ρυθμίσεις. Ίσως να είμαστε, θα έλεγα, στα όρια αυτού που θα ήθελε ένας μη Ευρωπαίος επενδυτής, αλλά έχουμε το πρόβλημα το ότι έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι εχθρική στην τεχνολογία και στον κίνδυνο. Τέλος, θα ήθελε η Κομισιόν να κάνει μια πραγματική μελέτη αντικτύπου για το τι θα σήμαινε αυτό η κάθε πιθανότητα, ευκαιρίες και κίνδυνοι να τα ζυγίσει. το τι θα μπορούσε να γίνει με μια μικρορύθμιση των υφιστάμενων ρυθμίσεων, υφιστάμενων ρυθμίσεων και να προσπαθήσει να διασφαλίσει ε, το ότι θα έχουμε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Κανείς δεν θέλει ενιαίους φόρους, τουλάχιστον εγώ δεν θέλω, αλλά χρειαζόμαστε ένα πιο αξιόπιστο πλαίσιο. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον συγκρίσιμες καταστάσεις και να ελέγξουμε μήπως ειδικά για ε, μεγάλα έργα επενδύσεων έχουμε κάποια φορολογικά πλεονεκτήματα. να ευνοηθούν φορολογικά για να υπάρχει ένα κίνητρο. Αυτά σας ευχαριστώ, αναμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Για τους κοιόδης εισηγητές, Αλφρέντο Παλώνη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Βόλφα για την εξαιρετική εργασία που έχει κάνει και πέρα από την εργασία του αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα περισσότερο και για την διαλλακτικότητα την οποία είχε στις επαφές που είχε μαζί μας για ένα ζήτημα το οποίο πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την στρατηγική ανάπτυξη, οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν λοιπόν πολύ ανοιχτό, πολύ διαλλακτικό και θεωρώ πραγματικά ότι μπορούμε να κινηθούμε αυτή τη στιγμή από κοινού και ότι συμφωνούμε τελικά για την ε, χρηματοδότηση αυτή τη μακροπρόθεσμη η οποία συνδέεται όλο και περισσότερο ως παράγοντας με την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να ασκήσουμε και μια κάποια κριτική. μόνο ότι συμφωνώ με την ε, γενικότερη στάση που έχει τηρηθεί μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι έχουν μειωθεί πάρα πολλοί επενδύσεις εξαιτία της κρίσης και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για αυτό το λόγο έχουμε και μία κρίση όσον αφορά την ίδια την απασχόληση. Ένα 75% των εταιριών μας εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τον τραπεζικό τομέα καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια ιδιαιτερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλε περιοχέ του κόσμου όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει ένα υψηλότατο επίπεδο εξάρτηση των επιχειρήσεών μα και πλήττονται περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσει, οι οποίε δεν καταφέρνουν να έχουν τα απαραίτητα δάνεια τα οποία χρειάζονται για να κάνουν επενδύσει και για να αναπτυχθούν. Πρέπει λοιπόν να βρούμε του κατάλληλου τρόπου για να ξεκινήσουν νέε επενδύσει. Πρέπει να καταφέρουμε να κινηθούμε προ μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα αναπτύσσεται οικονομικά. Νομίζω ότι καταρχά θα πρέπει να ασχοληθούμε με του θεσμικού επενδυτέ και θα πρέπει στη συνέχεια να καταφέρουμε να βοηθήσουμε και του ίδιου του ιδιώτες, τα ίδια τα νοικοκυριά, να κάνουν μακροπρόθεσμε επενδύσει μέσω δανεισμού θα ήθελα να καταθέσω μια προσωπική παρατήρηση που νομίζω ότι ε, συμφωνείς και εσύ με αυτήν, Βόλφ. Δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε μόνο στο πρόβλημα που υπάρχει με την ε, ανάληψη κινδύνου. Πιστεύω ότι υπάρχει και ένα πολιτιστικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες δεν επιθυμούν να κάνουν επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε και μία συζήτηση όσον αφορά το ζήτημα της φορολογίας, να πετύχουμε μία κάποια ευρωπαϊκή εναρμόνιση. Γιατί αυτό συνδέεται και με τη συζήτηση που κάνουμε πριν από λίγο. Η εναρμόνιση στην ευρωπαϊκή φορολογία, μια ευρωπαϊκή εναρμόνιση στη φορολογία μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε καλύτερες επιλογές όσον αφορά το οικονομικό περιβάλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι πέρα από τις επενδύσεις θα πρέπει να καταφέρουμε να καταστήσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ελκυστική όσον αφορά τους ξένους επενδυτές. Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός δρόμος για να καταφέρουμε να φτάσουμε στην οικονομική ανάκαμψη. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλοι θέλουν μια πιο φιλελεύθερη προσέγγιση, άλλοι μια πιο αντικυκλική προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μοναδική λύση η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί αμέσως. Επί του παρόντος, νομίζω ότι χρειαζόμαστε κυρίως περισσότερη Ευρώπη οι ευρωβουλευτέ αλλά και οι βουλευτέ από τη χώρα μου, την Ιταλία, λένε αυτό ακριβώ το πράγμα. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό το, πράγμα. Περισσότερη αλληλεγγύη αλλά και καλύτερη ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα από του δημοσιονομικού κανόνε, χρειαζόμαστε και κανόνε και ένα διάλογο για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Οι ε, τροπολογίε μου θα κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντω σα λέω ευθύ εξ αρχή ότι συμφωνώ με την πρώτη παρουσίαση που μα έκανε ο συνάδελφο Βόλφ. Νομίζω ότι οι απόψει μα για περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη Ευρώπη συγκλίνουν. Χρειαζόμαστε πέρα από μια οικονομική Ευρώπη και μια Ευρώπη των λαών και μια Ευρώπη αλληλεγγύη. Για ε, Σε ευχαριστώ, Σάρον. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βόλφ που έχει κάνει για το ζήτημα αυτό. Η συμβολή του αποτελεί πραγματικά μια καταπληκτική βάση εργασία, την οποία εμεί θα πρέπει κάπω να συμπληρώσουμε. Η πράσινη βίβλο Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα προτείνει κάποιε πλατφόρμες που θα μπορούσαμε εμεί να εκμεταλλευτούμε περισσότερο όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, σε ένα πλαίσιο όμω, ένα περιβάλλον, το οποίο επηρεάζεται πάρα πολύ από την μακροοικονομική κρίση και όπως καταλαβαίνετε είναι ο τομέας των επενδύσεων, αυτός ο οποίος παρουσιάζει πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Οι δημόσιες επενδύσεις είναι μόνο 2% σε σχέση με τα υψηλά ποσοστά που είχαμε στο παρελθόν και 17% τώρα σε σχέση με 28% το 2007. Όσον αφορά την πρόταση του εισηγητή για να υποστηρίξουμε περισσότερο τις αναπτυξιακές τράπεζες. Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή είναι θετική. Πρέπει ωστόσο να συμπεριλάβουμε στην έκθεση αυτή την έννοια του μακροπρόθεσμου δημόσιου επενδυτή, έννοια η οποία υπάρχει σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία για παράδειγμα. Θέλουμε περισσότερο επενδυτές που θα εντάσσονται περισσότερο στον τομέα αυτό και όχι τόσο πολύ να επιμένουμε στο ζήτημα των δημοσίων τραπεζών ανάπτυξης. Νομίζω ότι οι δημόσιοι αυτοί οι επενδυτές στους οποίους αναφέρομαι μπορούμε, μπορούν να υποστηρίξουν τόσο, την δημόσια, όσο, τόσο τις δημόσιες όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Πιστεύω, όπως λέγεται άλλωστε και στο άρθρο 8 της έκθεσης, ότι θα πρέπει να στηριχτούμε κυρίως στις τράπεζες, ότι οι τράπεζες θα πρέπει να, αποτελέσουν, να αποτελέσουν τη βασική μορφή χρηματοδότησης, Ωστόσο, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε τους μακροπρόθεσμους επενδυτές προκειμένου να συμβάλλουν μακροπρόθεσμα τελικά στην οικονομική ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να καταφέρουμε να προσαρμόσουμε αναλόγως τους προληπτικούς κανόνες και τους λογιστικούς κανόνες. Ο συνάδελφος Παλώνε, καθώς επίσης και ο Βόλφ, αναφέρθηκαν στο ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια νομική βεβαιότητα και σταθερότητα για τους επενδυτές. Επ' αυτού συμφωνούμε προφανώς, αλλά διαφωνούμε κάπως ως προς τον τρόπο που θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Συμφωνώ περισσότερο με τον κύριο Παλώνε, αν θέλετε. Μέσω μιας φορολογικής εναρμόνισης μπορούμε να το πετύχουμε αυτό περισσότερο. Και όντως ακολουθώντας τις προτάσεις του κυρίου Παλώνε μπορούμε να καταλήξουμε όντως σε κάτι τέτοιο. Νομίζω επίσης ότι θα ήταν θετικό, όπως το είπε και ο ίδιος ο εισηγητής, να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να καταφέρουμε να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβασή τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο έχει να κάνει με την τίτλοποίηση. η ε, διαδικασία εξυγίανσης των ισολογισμών των τραπεζικών ε, συνεχίζεται στη διαδικασία σε πολλές χώρες με την εξαίρεση κάποιων χωρών. Συνεχίζουν οι τράπεζες να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Σε καμία περίπτωση θα πρέπει όμως να θέσουμε μέσω της έκθεσης αυτής στην αμφιβόλο την πρόοδο που είχε επιτευχθεί από το 2009 και μετά όσον αφορά την, ε, τη ρύθμιση των τραπεζών. Εγώ σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν μετανιώνω για την εργασία που έχουμε κάνει για την οδηγία περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η εργασία του συναδέλφου Κάρα ήταν πάρα πολύ σημαντική και πολλοί οικονομολόγοι φοβούνται ότι ε, η τιτλοποίηση αποτελούσε ανέκαθεν έναν τρόπο για να παρακάμψουμε τους κανόνες της Βασιλείας Τρία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί Ας υπενθυμίσουμε ότι μέσω της τιτλοποίησης καταλήξαμε στην κρίση των ανυπόθηκων πιστώσεων υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ, καθώς επίσης και σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ας μην ξεχνάμε ότι μέσω της τιτλοποίησης πολύ συχνά διαχέουμε τοξικά προϊόντα στην αγορά παράγωγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Επομένως, είναι επόμενο στη συνέχεια στους ισολογισμούς των τραπεζών να βρίσκουμε και τα προϊόντα αυτά τα τοξικά. Ας είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί στις αναφορές που κάνουμε στην τιτλοποίηση. Χρειαζόμαστε, όπως το είπε και ο Βόλφ, τιτλοποίηση πολύ υψηλού επίπεδου, υψηλής ποιότητος. Πρέπει λοιπόν να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να δούμε τελικά τι είναι αυτή η τιτλοποίηση υψηλού επίπεδου, υψηλής ποιότητος. Πολύ ενδιαφέρουσα η έννοια αυτή αλλά θα πρέπει πραγματικά να είμαστε όλοι σύμφωνοι για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για τιτλοποίηση στοιχείων ενεργετικού υψηλή ποιότητα. Επίση, πρέπει να έχουμε κοινά πρότυπα όσον αφορά τι υπεύθυνε επενδύσει, να καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να επιμείνουμε περισσότερο στην δέουσα, σωστή, κοινωνική και περιβαλλοντική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, προκειμένου να μην δώσει απλώς λευκή επιταγή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σημείο αυτό. Θα καταθέσω λοιπόν τροπολογίες οι οποίες θα συνάδουν με τα όσα σας είπα και προσβλέπω σε μια πολύ επικοδομητική συνεργασία με τον εισηγητή και με τους πιο εισηγητές για τα σημαντικότατα αυτά ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Now for the Greens, uh, I have Bass down, but it doesn't look like it's going to be Bass. <laughs> τον Μπάς έχω σημειώσει εγώ για τους πράσινους, αλλά δεν μου μοιάζεται πολύ με τον Μπάς. Ναι, ε, ε, ο ο συνάδελφος ε, Μπάσε Κούτ ε, που είναι αρμόδιος στην ομάδα Πρασίνων για αυτό το ζήτημα. Έχει ένα κόλλημα και δεν ε, μπορέσει να παρευρεθεί, αλλά θα έρθει σε άμεση επαφή με τον εισηγητή. Ήδη γνωρίζει πολύ καλά το περιεχόμενο του σχεδίου. Ευχαριστώ από τους συντηρητικούς. Ένας άλλος, κάποιος άλλος ε, πάλι αντικαταστάτησε, έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι εγώ σκιώδης βεβαίως, είναι η κυρία Βόρντεντ, όπως ε, καταλαβαίνετε. Ε, προετοιμάζει βεβαίως κάποιες τροπολογίες. Άκουσα τον κύριο Κλίντς πολύ προσεκτικά, έχω κάποιες παρατηρήσεις. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα πως η έκθεση αυτή θα είναι λογική και βεβαίως ε, οι απόψεις μας ε, διαφέρουν ε, για το πώς θα ξεκινήσει η οικονομική ανάπτυξη, πώς θα δώσουμε ένα κίνητρο στην ανάπτυξη. Οπωσδήποτε διαφέρουμε και βεβαίως δυστυχώς ο κύριος Λάμπερτς ε, δεν είναι εδώ. Μπορούμε να συνεχίσουμε την ε, συζήτηση, αλλά ε, πρώτα απ' όλα κάποιες παρατηρήσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Κλίντς όταν λέει πως ε, χρειάζεται ένα σταθερό και διάφανο αριθμιστικό πλαίσιο για εμένα το ερώτημα είναι το εάν ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Κοιτάξτε, συζητάμε το ρυθμιστικό πλαίσιο εδώ και χρόνια και υπάρχουν πάρα πολλοί κανονισμοί που καθιστούν τελικά το σύστημα λιγότερο κατανοητό και διάφανο. Μήπως οι πάρα πολλοί κανονισμοί περιορίζουν την ανάπτυξη. Αυτό θα έλεγα εγώ. Δεύτερον, μία συζητήσιμη παρατήρηση. Αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε για ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αλλά θα ήμουν πιο προσεκτικός γιατί Εγώ επειδή είμαι υπέρ του φορολογικού ανταγωνισμού, δεν ξέρω αν θα ήμουν υπέρ του συντονισμού των φορολογικών πολιτικών. Αυτό έτσι παρανθετικά για αυτό το οποίο είπε πριν από λίγα λεπτά ο κύριος ε, Λαμπέρτς. Πολύ απλά λειτουργεί ο φορολογικός ανταγωνισμός. Και πρέπει να τον αφήσουμε να λειτουργήσει. Λοιπόν, αυτές οι παρατηρήσεις από μένα δεν είμαι σκιώδης ηγητής. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει γκουε. Οπότε περνάμε στους λοιπούς ομιλητές. Ευχαριστώ. Δύο-τρει σύντομε παρατηρήσει ε, για την ανάλυση. Ε, θα συμφωνήσω με τον Βόλφ Ε, στο μόνο με το οποίο θα διαφωνήσω μαζί του και θα συμφωνήσω με τον Αλφρέντο και τον Λίμε είναι το ζήτημα τη φορολογική ε, διαχείριση. Δεν μπορούμε να λύσουμε με αποτελεσματικό τρόπο το ζήτημα τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση παρά μόνο με εναρμόνιση φορολογικών βάσεων και μια λογική εναρμόνιση των συντελεστών. Αλλιώ θα έχουμε έχουμε πάντα φορολογικό ανταγωνισμό. Ε, για την τυκλοποίηση θα συμφωνήσω με τον Βόλφ. Ε, χρειαζόμαστε τυπλοποίηση υψηλής ποιότητας, ε, αλλά σίγουρα είναι απαραίτητη η τυκλοποίηση για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ως ε, μοναδικό σημείο αναφορά στην ενυπόθηκα δάνεια τα subprimes. Στατιστικά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι παρότι υπήρξαν μεγάλες αποτυχίες και χρεοκοπίες ε, στη ΣΥΠΑ λόγω των λοιπόν η ευρωπαϊκή τιτλοποίηση ε, ε, είχε πολύ πιο σοβαρά αποτελέσματα διότι δεν περιείχε τέτοια ενυπόθηκα. Οπότε ε, για τη μακροπρόθεσμη νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε την τιτλοποίηση. Ευχαριστούμε η Ίντα. Γκάλπελτς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά βάση συμφωνώ με τις παρατηρήσεις ε, του κυρίου Κλίντς, αλλά θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Όσον αφορά το σημείο 5, πρώτα απ' όλα, είναι γεγονός πως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τράπεζες παρέχουν την ε, περισσότερη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Αλλά αυτό δεν είναι αποτέλεσμα κακής διαχείρισης ε, κάποιας δημόσιας διοίκησης, οπωσδήποτε οι επενδύσεις πρέπει να είναι ασφαλείς ε, και διαφανείς. Είναι σημαντικό αυτό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αλλά όσον αφορά τις νέες ε, πηγές χρηματοδότησης, πρέπει να τονίσουμε τον ρόλο των ε, κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά τις μελλοντικέ ε, δυνατότητες ε, χρηματοδότησης. Δεν συμφωνώ πως το κράτος είναι αξιωματικά κακός διαχειριστής ή διοκτήτης. Επίσης συμφωνώ πως είναι καλή ιδέα να δημιουργηθούν τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες. Αυτό θα είναι θετικό ειδικά για διασυνοριακά έργα. Περιφερειακές ε, τέτοιες τράπεζες λοιπόν θα είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Το, το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να διευκολύνει τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά πρέπει να σημειώσουμε πως ε, η ενιαίες διατάξεις ε, για την ε, λογιστική βεβαίως θα ενισχύσουν την ε, λογοδοσία και την διαφάνεια. Τέλος, για, για την εναρμόνιση της φορολογίας και τις φοροαπαλλαγές κτλ. Κοιτάξτε, βραχυπρόθεσμα η εναρμόνιση φορολογίας δεν είναι σωστή απάντηση στα προβλήματα των έργων υποδομών νομίζω πως ε, μπορούμε να μιλήσουμε για φορολογική εναρμόνιση το πολύ πολύ ε, μακροπρόθεσμα. Ίσως το μέλλον να είναι μια καλή ιδέα, αλλά αυτή τη στιγμή ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τον συντονισμό. Σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Όχι. Βολφ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλια. Καθώς και εκείνους που αντικατέστησαν τους σκιώδεις που δεν είναι εδώ σήμερα, κάποιες απαντήσεις να δώσω. Όταν λέω ότι χρειαζόμαστε ένα σταθερό περιβάλλον, δεν αναφέρομαι αναγκαστικά σε πλήρη εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών. Θέλουμε απλώς ένα σύστημα το οποίο να μην τροποποιείται πάρα πολύ από τον ένα στο άλλο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Αλιαντς, η μεγαλύτερη γερμανική ασφαλιστική εταιρεία, έκανε μία μακροπρόθεσμη επένδυση στην Ορβηγία, γιατί από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ υγιής η επένδυση αυτή. Δύο χρόνια μετά την έναρξη της επένδυσης αυτής, άλλαξε το φορολογικό καθεστώς στην Ορβηγία σε τέτοιο βαθμό που τελικά ε, μειώθηκε κατά το ίμιση οποιαδήποτε δυνατότητα κέρδους από την επένδυση αυτή και καταλαβαίνετε ότι αυτό λειτουργεί πάρα πολύ αποθαρρυντικά για τις ξένες άμεσες επενδύσεις. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ένα σταθερό περιβάλλον, όπως σας είπα, σε αυτό αναφερόμουν. Ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάω μια στιγμή το χρονοδιάγραμμά μας. 3 Δεκεμβρίου το μεσημέρι είναι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και θα συζητήσουμε την συζήτηση αυτή στις 9 Ιανουαρίου και θα ψηφίσουμε στις 22 Ιανουαρίου στην Επιτροπή και θα περάσει η έκθεση στη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Έχουμε καταφέρει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό λίγο νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν στη ημερήσια διάταξη. Σας προτείνω να κάνουμε ένα σύντομο πεντάλεπτο διάλειμμα, έτσι ώστε να δούμε ότι όλοι έχουν έρθει όσοι πρέπει να βρίσκονται εδώ πέρα και ξεκινάμε πάλι, συνεχίζουμε μάλλον την συνεδρίασή μας σε πέντα λεπτά. Αυτά όσον αφορά το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή την οικονομική συμμετοχή των υπαλλήλων στα εταιρικά έσοδα. Okay. Ah, the rapporteur. Oh, yeah, he's there. He's walking back Just to his checking place. we've got everybody back again. Θέλω να δω αν είμαστε όλοι στην αίθουσα, αν δεν έφυγε κανείς στο διάλειμμα. Ας περάσουμε λοιπόν στο σημείο 6 της σημερίσιας διάταξης. Έκθεση από τον Φαμπρίτσιο Μπερτό Εξέταση τροπολογιών όσον αφορά την οικονομική συμμετοχή των υπαλλήλων στα εταιρικά έσοδα. Ο συγητής έχει το λόγο. Τόσο παρέμβαση. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έλεγα ότι εργάστηκα για την σύνταξη της έκθεσης αυτής που είχα και τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω πριν από μερικές εβδομάδες στην Επιτροπή μας και έχω λάβει 28 τροπολογίες. Θα έλεγα μία τροπολογία για κάθε φράση της έκθεσής μου. Συνεργάστηκα λοιπόν με τους κοιόδης εισηγητές, με όλους τους συμβούλους από όλες τις πολιτικές ομάδες, προκειμένου να καταφέρω να περιορίσω τον αριθμό των τροπολογιών και προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάποιες ε, συμβαστικές τροπολογίες. Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στα ερικά έσοδα και αυτή η συμμετοχή να αποτελέσει τελικά χρηματοδότηση των ίδιων των εταιριών. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να γίνουν και κάποιες αναφορές στην φορολογική πολιτική των κρατών μελών και όπως ξέρετε δεν έχουμε εμεί άμεση αρμοδιότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη και τις εταιρείε. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε απλώς κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Θα έλεγα όμω ότι γενικόταν και το κείμενο της καθήλυνα αρμόδια επιτροπής, τη Επιτροπής Απασχόλησης δηλαδή. Θα ακούσουμε φαντάζομαι και του συντάκτε των τροπολογιών για τις μέρου τροπολογίες. Απλώ να πω εγώ ότι από τις 28, αυτέ τροπολογίε αυτές οι περισσότερες είναι αποδεκτές. Εφόσον τελικά είναι τροπολογίε που βελτιώνουν το αρχικό δικό μου κείμενο και ουσιαστικά κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με αυτή την οποία σας εξέθεσα στην πρώτη παρουσίαση της γνωμοδότησης. Επίσης, όπως σας είπα, έχουμε καταλήξει και σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες, εκ των οποίων δύο από τις τρεις έχουν τη σύμφωνη γνώμη των συντακτών τροπολογιών. Υπάρχει απλώς ένα προβληματικό σημείο που νομίζω τελικά και πέρα θα επικεντρωθούμε σήμερα στη συζήτησή μας. Το σημείο αυτό λοιπόν που έχει να κάνει με τη λεγόμενη τροπολογία B, Β μέσω της οποίας θέλουμε τελικά να αναφερθούμε στην δυνατότητα ορισμένων εργαζομένων οι οποίοι για οικονομικούς λόγους έχουν αποκλειστεί από τη δραστηριότητα της επιχείρησης, δηλαδή άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους, τον οποίο τερματίστηκε η σύμβαση για οικονομικούς λόγους, μπορούν, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί μέσω των αποταμιεύσεών τους ή μέσω των ε, επιδομάτων ανεργίας ή μέσω άλλων κοινωνικών επιδομάτων που λαμβάνουν να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί μετά από δική τους προφανώς επιλογή και με την ε, σύμφωνη γνώμη της ίδιας εταιρεία να μπορούν να συμβάλλουν οι άνθρωποι αυτοί στη χρηματοδότηση της ίδιας εταιρεία, και θα μπορούσε σε αντάλλαγμα εταιρεία να τους ξαναπροσλάβει. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα εντάσσονται εκ νέου στον παραγωγικό κύκλο και θα μπορούσαν κατά αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι αυτοί να διατηρήσουν τη θέση απασχόλησής τους μέσα στην εταιρεία στην οποία εργαζόντουσαν στο παρελθόν. Θα καλούσα όλους τους συναδέλφους που δεν συμφωνούν με την πρόταση αυτή, με την τροπολογία αυτή τη συμβαστική, να το σκεφτούν λίγο ακόμα. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μέτρο αυτό είναι καθαρά κοινωνικό μέτρο τελικά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο κοινωνικό από το να μπορεί κανείς να υποστηρίζει έναν εργαζόμενο, να υποστηρίζει την αξιοπρέπεια ενός εργαζομένου. Και νομίζω ότι είναι και απολύτως φιλελεύθερο από την άλλη. Χρησιμοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο δημόσιοι πόροι, οι οποίοι θα δαπανώνταν διαφορετικά. Χρησιμοποιούνται οι δημόσιοι αυτοί πόροι, για παράδειγμα τα επιδόματα ανεργίας, με έναν τρόπο καθαρά αποδοτικό παραγωγικό. Ουσιαστικά τα επιδόματα αυτά ανεργίας ή αποταμίευση των εργαζομένων συμβάλλει στην ε, ίδια τη χρηματοδότηση εταιρεία, η οποία με τη σειρά τη μπορεί να επαναπασχολήσει του εργαζομένου αυτού. Πρόεδρο, σα ευχαριστούμε πολύ. Μόικα Κλέβα για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή για την έκθεση και για τις τρεις προτινόμενες συμβαστικές τροπολογίες. Έχουμε ένα καλό κείμενο εδώ πέρα που βεβαίως συμπεριλαμβάνει τις θετικές τάσεις που βλέπουμε σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Επίσης θεωρώ πως το θέμα αυτό, ειδικά σε καιρούς που προσπαθούμε να αντιπαλέψουμε τις αιτίε και συνέπειες της κρίσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό ένα βασικό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα βοηθήσει τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές ε, πρέπει να στηριχθεί. Θεωρώ λοιπόν ε, ότι ένα σύστημα αμοιβαία αναγνώρισης τέτοιων συστημάτων στην Ευρώπη ε, πρέπει να αρκεί. Δεν χρειάζεται περισσότερο να παρέμβει η Κομισιόν. Επίσης πρέπει να εστιαστούμε σε μακροπρόθεσμο όραμα, να είναι σε θελοντική βάση και βεβαίω να ακολουθεί ε, τις αρχές συμμετοχής των εργαζομένων και τις ε, σε επιμέλης. Όσον αφορά τώρα τη φορολογική πολιτική, ε, υπάρχει αρκετά μεγάλο περιθώριο ελιγμών θα έλεγα και ταυτόχρονα δουλειά που πρέπει να γίνει. Οπωσδήποτε θα ζητούσα από την Κομισιόν να εξετάσει το ζήτημα αυτό, να, μαζέψει, να βρει κάποια παραδείγματα ειδικά βέλτιστων πρακτικών και να καθορίσει κάποιες βασικές ευρωπαϊκές αρχές για τις σχέσεις αυτές. Τέλος, οπωσδήποτε συμφωνώ πως πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος στο ζήτημα το φορολογικό, ειδικά το πρόβλημα της πιθανής διπλής φορολογίας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βρεθεί ένας ευρωπαϊκός τρόπος να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές ε, στο σχεδιασμό και προσανατολισμό ε, φορολογικών ε, οφελών και κινήτρων. Επίσης, αν μου επιτρέπετε, είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα, αλλά έχω κάποια προβλήματα ως προς την εφαρμογή. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από τους άλλους συναδέλφους να κάνουν κάποιες προτάσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο για να το στηρίξει και η ομάδα των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για την άλλη ο Φιλίπ Ντεμπάκερ λείπει. Θα μιλήσει κάποιος θέση του. Όχι. Για τους πράσινους. Α, ο Φιλίπ. Έλα. Πάνω στην ώρα. Ναι, ναι, έχουμε προχωρήσει. έτσι ευέλικτη φιλελεύθερη. Λοιπόν, όταν είσαι έτοιμος έχεις το λόγο. Λοιπόν, βεβαίω ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει και για τις συζητήσεις που είχαμε. Πάντα είχαμε τις ίδιες αρχές, ότι είναι σημαντικό δηλαδή η οι υπάλληλοι να έχουν κίνητρο να μην στην εταιρεία, αλλά και κάποιο άλλο κίνητρο, αυτό της οικονομικής συμμετοχής. Ε, τέτοια στήματα υπάρχουν ήδη σε πολλές εταιρείες προαιρετικά. Πρέπει λοιπόν να έχουν την επιλογή οι υπάλληλοι και οι εταιρείε ε, για τέτοια στήματα και το πώς θα τα διαμορφώσουν. Για τις συμβαστικές προτάσεις ε, ε, συμβαστική τροπολογία 1 συμφωνούμε με τη φιλοσοφία του κειμένου, αλλά προσπαθούμε να πούμε το ίδιο πράγμα δύο-τρει φορέ. Οπότε, ίσω θα μπορούσαμε να ζητήσουμε κάποια αναδιατύπωση, Χωρί να αλλάξει τίποτα στην ουσία. Απλά επειδή η ίδια πρόταση επαναλαμβάνεται στην αρχή και στο τέλο παραγράφου να διαγραφεί. Συμβαστική τροπολογία Γ και αυτή μπορούμε να τη στηρίξουμε. Σαφής ε, τροπολογία και απλά δήλωση των γεγονότων. Ε, με την Β βεβαίως έχουμε ένα ζήτημα, δηλαδή ε, αν ε, φύγουν από μια εταιρεία οι εργαζόμενοι μπορούν να επενδύσουν αλλού, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τους άλλους μετόχους, γιατί είναι πλέον μέτοχοι. Οπότε η πρόταση που έχετε κάνει δεν προσθέτει κάτι, δεν τους εμποδίζει δηλαδή σήμερα κάτι να το κάνουν αυτό. Οπότε για εμάς η συμβαστική Β είναι κάτι το δύσκολο. Αυτά εν ολίγης ε, είναι η άποψή μας. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη που θα σας να προφανώς το λόγο, απλώς δεν ήσασταν στην αίθουσα και πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα από τους πρασίνους, κανείς, από τους συντηρητικού, από το ECR. Ο Σάικα αλλά δεν είναι εδώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο και πάλι θα τελειώσουμε το σημείο αυτό πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, δεν υπάρχουν ε, άλλοι ομιλητέ, επομένω δίνω πάλι το λόγο στον, συντάκτη γνωμοδότηση. Φαμπρίτσιο, έχει το λόγο. Σε σχέση με την άποψη της Άλντε, έχω λάβει εδώ πέρα μία ανακοίνωση, μία πληροφορία που έχει να κάνει με τη συμβαστική τροπολογία Β από ό,τι φαίνεται, θα μπορούσατε να υπερψηφίσετε την τροπολογία αυτή αν τη χωρίζαμε σε επιμέρους τμήματα. Όσον αφορά εμένα, μπορούμε να χωρίσουμε σε τμήματα την τροπολογία αυτή. Δεν έχω κάποια αντίρρηση. Άρα μπορείτε κι εσείς να ταχτείτε ευνοϊκά υπέρ της τροπολογίας αυτής, έτσι δεν είναι της συμβαστικής τροπολογίας Β. Να απαντήσω προφανώ, λέει ο κύριο Δεμπάκερ. Νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση εδώ πέρα. Η όλη ιδέα πίσω από την τροπολογία Β, ότι κάποιο ο οποίο απολύεται μπορεί να επενδύσει τα χρήματά του στην εταιρεία αυτή και ότι η εταιρεία θα έχει μετά την υποχρέωση να τον ξαναπροσλάβει, είναι κάπω περίεργο σαν έννοια για μένα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι Έχουμε εδώ πέρα δύο, τρία μάλλον, τρεις διαφορετικές σχέσεις μπορούμε να έχουμε μια εταιρεία. Την καθαρά εργασιακή σχέση, αλλά και τις σχέσεις οι οποίες προκύπτουν από τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο. Θα είναι σαν να λέμε μέσω της τροπολογίας αυτής ότι ε, η εταιρεία έχει την υποχρέωση να προσλάβει ως εργαζόμενους όλους τους μετόχους της. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε εμείς τέτοια υποχρέωση η επιχείρηση είναι αυτή η οποία αποφασίζει τελικά για το ποιο θα προσλάβει και ποιο όχι. Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε εμεί να υποστηρίξουμε την τροπολογία αυτή, ιδίω με τον τρόπο που διατυπώνεται. Και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ακόμα και αν χωρίσουμε την τροπολογία αυτή σε επιμέρου τμήματα. Όπω σα είπα, δεν βλέπω ποια είναι η προστιθέμενη αξία πίσω από αυτή την τροπολογία. Πρόεδρο, θέλει να απαντήσει ο εισηγητή. Και αν δεν κάνω λάθο, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να πάρει το λόγο. Όντως έχουμε αρκετό χρόνο στην ε, διάθεσή μας, γιατί θα καθυστερήσει ο εισηγητής ε, του επόμενου σημείου της ημερήσιας διάταξης. Μόνος μπορούμε να το απολαύσουμε, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Μπερτό. Κοιτάξτε, δεν θέλω απλώς να γεμίσω τώρα το χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας. Να πω πάντως ότι ε, Εγώ άκουσα προσεκτικά τον κύριο Ντεμπέκερ, πάντως έχω μπροστά μου ένα έγγραφο από τους αφιλελευθέρους, το οποίο ζητά έναν χωρισμό σε τμήματα της συμβαστικής τροπολογίας Β. Και αυτό το που είπα εγώ είναι ότι θα συμφωνούσα με ένα τέτοιο διαχωρισμό της τροπολογίας σε τμήματα, αν αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ταχθεί η άλντε υπέρ της τροπολογίας αυτής. Τώρα, η, ε, όλη αυτή η θεωρία ότι θα πρέπει όσοι χρηματοδοτούν μια εταιρεία μέσω συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο να αντιμετωπίζονται με ισότιμο τρόπο είναι, κοιτάξτε, μια πρόταση που έχει να κάνει κυρίως με την υφιστάμενη περίοδο οικονομικής κρίσης ουσιαστικά εδώ πέρα αναφερόμαστε στο ζήτημα περισσότερο της απασχόλησης και ότι θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις από τα κράτη-μέλη στην απασχόληση. Ουσιαστικά θέλουμε εδώ πέρα να προωθήσουμε μία επένδυση δημοσίων πόρων προς μια εταιρεία. Πρόκειται για πόρους που με τη μορφή επιδομάτων ανεργίας δίνει ένα κράτος, δίνει το δημόσιο προς έναν άνεργο. Έλεγα λοιπόν ότι θα μπορούσε ο άνεργος αυτός να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να επενδύσει στην εταιρεία που τον απέλησε και η εταιρεία αυτή θα είχε την υποχρέωση να τον επαναπροσλάβει. Θα μπορούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο να αξιοποιήσουμε καλύτερα κάποιους πόρους. Ξέρετε ότι η συγκεκριμένοι αυτή πόροι, τα επιδόματα ανεργίας, ουσιαστικά πηγαίνουν μόνο στους ανέργους. Μέσω λοιπόν της τροπολογίας αυτής θα μπορούσαμε να εξοπλίσουμε καλύτερα τους δημόσιους αυτούς πόρους, εν προκειμένου τα επιδόματα ενεργείας, για να χρηματοδοτηθεί μια επιχείρηση, μια εταιρεία. Δεν κάνουμε λοιπόν εμεί τη διάκριση αυτή, στην τροπολογία αυτή. Η διάκριση αυτή υπάρχει ούτω ή άλλω όσον αφορά του δημόσιου αυτού πόρου. Τώρα, όσον αφορά τι παρατηρήσει από του σοσιαλιστέ, μπορώ να πω ότι συμφωνώ μαζί του. θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περισσότερο μέχρι αύριο που θα ψηφίσουμε για την γνωμοδότηση αυτή για να καταφέρουμε να πετύχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο συμφωνίας και σύγκλησης απόψεων. Πάντως, το κείμενο αυτό, το είπαν οι ακολουθεί μια φιλοευρωπαϊκή πορεία. Και ουσιαστικά στόχος του κειμένου επίσης είναι να εντοπίσει καλύτερα τις ε, ευκαιρίες χρηματοδότησης ε, για μία εταιρεία και για το πώς θα μπορούσαν τελικά οι ίδιοι εργαζόμενοι να συνδεθούν περισσότερο με την εταιρεία τους μέσω συμμετοχής τους στα εταιρικά έσοδα της επιχείρησης αυτής. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σημεία σύγκλησης με τους ε, σοσιαλιστές και αυτό φαίνεται και από τα ίδια τα νούμερα. Όπως σας είπα, έχουν απορριφθεί δύο μόνο τροπολογίες από τις 28 που έχουν υποβληθεί. Επί τους ουσίας, λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνένεση όσον αφορά δηλαδή τις βασικές προτάσεις που πρέπει να υποβάλουμε προς την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Βέβαια, πρέπει να πω προς τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, ε, προς τον εκπρόσωπο μάλλον των Σοσιαλιστών, ότι η Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει ακόμα να καταβάλει πολύ σημαντικές προσπάθειες, προκειμένου να συμπληρωθεί ακόμα περισσότερο η έκθεσή τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, έχουμε ξεφύγει λίγο ε, χρονικά, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος πάντων, έχουμε 25 λεπτά μέχρι να έρθει ο επόμενος εισηγητής. Ε, και ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Αλλαγή ε, μπορεί να είμαι και γενναιόδορη, μπορώ να σας δώσω πολύ χρόνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θέλω να τονίσω ποιες δραστηριότητες έχει αναλάβει σε αυτό το τομέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, αυτό το ζήτημα συμπεριλήφθηκε στο σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εταιρική διακυβέρνηση και το εταιρικό δίκαιο που δημοσιεύσαμε πριν από ένα χρόνο ε, και τονίσαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό από οικονομική άποψη ε, να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα κέρδη τη εταιρεία ε, για την ενίσχυση τη διαφάνεια, την πρόθεση τη ποιότητα στην εταιρική διακυβέρνηση και μέσω της συμμετοχής τους στα κέντρα της εταιρεία ε, μέσω διαφόρων συστημάτων. Βάσει διαφόρων μελέτων βλέπουμε ότι αυτό ενισχύει βάρο πολύ την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αφενός και αφετέρου τα κίνητρα και την ε, ε, θετική συμμετοχή και συμπεριφορά των εργαζομένων. Αυτά έχουν θετικό αντίκτυπο της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Επίσης, αυτό συνδέεται άμεσα με το μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ίδιας εταιρείας, καθώς και τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας. Επίσης υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα του ε, Κοινοβουλίου για την, ε, συμμετοχή, ε, την αυξημένη συμμετοχή των εργαζομένων αξιολογηθούν τα σχετικά προγράμματα και τα ρυθμιστικά πλαίσια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αναλυθούν οι λόγοι για τον οποίο σημαίνονται αποκλήσει ω προς τι εθνικέ προσεγγίσει σε αυτό το ζήτημα ε, θα εξεταστούν οι των διαφόρων συστημάτων και θα εξεταστούν οι διάφορε νομοθετικέ και μη δράσεις που μπορούν να αναλυθούν το ώστε ε, να ε, αυξηθεί η οικονομική συμμετοχή ε, των εργαζομένων στις εταιρείε και να ενισχυθεί η γενικότερα η συμμετοχή τους. Θα εξεταστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο, το διοικητικό, το φορολογικό άχθος και ούτω καθεξής. Για τις βέλτιστες πρακτικές από τις διάφορες χώρες ε, θα, θα συζητηθεί το ζήτημα σε μια διάσκεψη που θα γίνει στις 30 ε, Ιανουαρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ με αυτή την ευκαιρία θα κάνει την εναρκτήρια ομιλία για να ε, υποστηρίξει την αυξημένη συμμετοχή των εργαζομένων στις εταιρείε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιος να επανέλθει ίσως, να δευτερολογήσει. Διαβουλεύεται ο εισηγητής μου. εσείς θέλετε, Φαμπρίτσιο. Ε, ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Μία απλή λεπτομέρεια θέλω να παραθέσω, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Μια λεπτομέρεια μόνο όσον αφορά την μετάφραση. Στο ιταλικό κείμενο, ο τίτλος της γνωμοδότησης αυτής αναφέρεται σε οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα έσοδα της εταιρείας στα κέρδη της εταιρείας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αντιστοιχεί στο λέξη profit στα αγγλικά, ενώ εμείς μιλάμε για την δραστηριότητα της επιχείρησης. Δεν θα ήθελα λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποιος Ιταλός, αν μη τι άλλο συνάδελφος, να φανταστεί ότι μιλάμε εδώ πέρα για τα κέρδη της εταιρείας. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην δραστηριότητα της εταιρείας, στη δραστηριότητα της επιχείρησης και όχι στα κέρδη της επιχείρησης. Πρόεδρος. Άλλος ομιλητής, όχι. Ο Ανδρέας Σουάπ θα καθυστερήσει 10 ε, λεπτά. Έχουμε λοιπόν 20 ε, λεπτά στην ε, διάθεσή μας και δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιο άλλο ζήτημα να συζητήσουμε στα 27 λεπτά. Θα κάνουμε λοιπόν ένα ακόμα σύντομο διάλειμμα για 15 λεπτά αυτή τη φορά και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ. Okay, everybody, we've captured our rapporteur. Λοιπόν, ήρθε και ο συγγητής, γιατί δεν ήταν εύκολο να έρθει. Οπότε, περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάση του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού εθνικής τε και κοινοτικής. Λοιπόν, ο εισηγητής είναι ο Ανδρέας Σφάμπ, ο οποίος έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι για το ότι σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για τις τροπολογίες. Την προηγούμενη εβδομάδα με τους χιώδης ήδη τα είπαμε και είχαμε ήδη μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με σημαντικά στοιχεία και ορίσαμε κάποιους στόχους. Επίσης χαίρομαι για το ότι συμφωνήσαμε ε, για το ότι η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού πρέπει να, να είναι ενιαία και αυτό είναι πρώτη προτεραιότητα για όλους. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προστατευόμενων μαρτύρων αλλά βεβαίως αυτό είναι μια περίπτωση ιδιαίτερος εξαιρετική. Επίσης ε, δεν ήταν δυνατόν βεβαίως να βρούμε συμβαστικές λύσεις ε, για όλα τα ζητήματα, αλλά νομίζω πως ε, η κυρία Νετφέλ θέλει να κάτσει και αυτή τη βδομάδα να τα ξαναπούμε, κυρίως για το ζήτημα του προγράμματος επί για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού. Χαίρομαι άρα για το ότι αύριο θα τα συζητήσουμε αυτά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν κυρία Πρόεδρε να σας δώσω μια γενική ιδέα για το που βρισκόμαστε γνωρίζετε. Πώς η Επιτροπή μας και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είχαν μια μικρή διαφωνία για το ποιος είναι υπεύθυνο για ποια ζητήματα και μετά από δύο μήνες επιτέλους συμφωνήσαμε και η Επιτροπή ε, Δικαίου είναι αρμόδια για, το, για τα άρθρα 5, 10, 17 και 18 και ε, βεβαίως ε, οι ορισμοί, συμπεριλαμβανωτικοί ορισμοί στο άρθρο 4 και τα αναλογα εκτιμώντας η Επιτροπή μας, κυρία Πρόεδρε, έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα άρθρα 6, 7, 9 και 19 μέχρι 22 και βεβαίως ε, το ανάλογο κομμάτι του άρθρου 4. Όλοι οι υπόλοιποι τομείς είναι κοινή αρμοδιότητα και βεβαίως έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Ράπκα, εισηγητή στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Βεβαίως δεν ξέρουμε πότε θα υποβάλει την έκθεση το δικό του σχέδιο έκθεσης και θα πρέπει να περιμένουμε άρα και την ψηφοφορία επί της δικής του έκθεσης και ανάλογα να προσαρμοστούμε. Όμως ελπίζω να μπορέσουν να ψηφίσουν στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων μέχρι τις 21 Ιανουαρίου και ε, μέχρι τότε να έχουμε και εμείς ε, υποβάλει τις ε, τροπολογίες μας έτσι ώστε 27 Ιανουαρίου να ψηφίσουμε και στην Επιτροπή μας. Στο Συμβούλιο θα τα έχετε ακούσει πως υπάρχει μια συζήτηση για τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για το εάν ε, το Συμβούλιο με βάση το άρθρο 103 είναι αποκλειστικά υπεύθυνο. Η Κομισιόν στηρίχθηκε σε δύο σημεία αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει να υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο για την αλλαγή της νομικής βάσης ε, και βεβαίως ε, υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για την επίτευξη αυτής της ομοφωνίας. Οπότε η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία και θα ήθελα να πω τα εξής υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες που υπέβαλα και εγώ. Γιατί, Γιατί το 10, ειδικά σε δύο περιπτώσεις, στην περίπτωση Ντόναου και μη, αλλά και σε μια άλλη απόφαση, είπε πως το απόρριτο εγγράφων που ζητάει η Κομισιόν σε περίπτωση προστατευόμενων μαρτύρων δεν μπορεί να αποτελέσει μια γενική περίπτωση. Και Μπορώ να πω ήδη πως η περίπτωση των ε, προστατευμένων μαρτύρων είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την προστασία των καταναλωτών γιατί πάρα πολλά καρτέλα δεν θα τα είχαμε ανακαλύψει καν χωρίς αυτούς τους μάρτυρες. Η σημαντικότερη ε, διαδικασία λοιπόν, οι σημαντικότερες διαδικασίες ε, τις οποίες έχει φέρει σε πέρας και ενώπιον του δικαστηρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετίζονται ακριβώς με τέτοιους μάρτυρες. Πρέπει λοιπόν και στο μέλλον να υπάρχει η διασφάλιση πως θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν αυτά τα προγράμματα και άλλοι μάρτυρες. Οπότε μπορούν οι επιχειρήσεις να ζητήσουν να μην τιμωρηθούν, αλλά δεν μπορούν να ζητήσουν να μην αποζημιωθούν οι πελάτες τους. Οπότε θα εξακολουθούν να είναι υπόχρεοι σε αποκατάσταση της ζημίας, αλλά βεβαίως μέσω της αυτοκαταγγελίας μπορούν α, κατά κανόνα να βρεθούν στην εξής κατάσταση ότι η εταιρεία η οποία θα καταγγείλει πρώτη το καρτέλ θα γλιτώσει την τιμωριακά το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζω λοιπόν πως ε, ε, έκανα μια αρκετά καλή εισαγωγή και αναμένω τώρα να δω τι θα πούν οι συνάδελφοι των άλλων ομάδων για τις ε, δικές τους τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay, thank you. Uh, now go to the shadow. Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε τώρα στους σκιώδεις ηγητές, πρώτα από τους σοσιαλιστές. Κύριο Σάντσετς, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σφάβ για την παρέμβασή του και βέβαια να τον ευχαριστήσω και για την πολύ καλή ανταλλαγή απόψε που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και παλιότερα. Προφανώς θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις. Το χρονοδιάγραμμα όμως μας πιέζει πάρα πολύ αν πραγματικά θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ. Όσον αφορά τη νομική βάση, να σας πω ότι όταν μιλάμε για το ζήτημα αυτό, ήταν ανέκαθεν σαφές ότι το ζήτημα αυτό έχει να κάνει με το δίκαιο ανταγωνισμού, αλλά έχει να κάνει επίσης και με την ευθύνη, με την αποτελεσματική ευθύνη, πράγμα το οποίο αποτελεί από μόνο του ένα πολύ σημαντικό τμήμα της νομικής βάσης. Ορισμένοι λοιπόν θεωρούν ότι θα πρέπει να προβλέπεται μια ξεχωριστή νομοθεσία για το ζήτημα το οποίο συζητάμε και γι' αυτό το λόγο η πρόταση που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νομική βάση μας δίνει τη δυνατότητα να επιτύχουμε τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε. Από τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, δύο μόνο θα καταπέσουν γιατί οι υπόλοιπες έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Εγώ έχω τις εξή ανησυχίε τώρα. Αναφερόμαστε εδώ πέρα στον πυλώνα ιδιωτικού δικαίου του ανταγωνιστικού δικαίου. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει το ζήτημα αυτό σε προηγούμενη παρουσίαση που έκανε και θυμάμαι τότε εκπρόσωποι των Σαριστών και του ΕΛΚ αναφέρθηκαν στο ότι θα πρέπει να δοθεί μια νομοθετική προτεραιότητα στο ζήτημα αυτό, ιδίω όσον αφορά την συλλογική προσφυγή, τους μηχανισμούς συλλογικής ένομης προστασίας. Το σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν αναφερόμαστε εδώ πέρα μόνο σε συλλογική προσφυγή, αλλά γενικότερα σε προσφυγές. Η βασική αρμοδιότητα, όπως γνωρίζετε, είναι αυτή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και ελπίζω ότι θα κρατήσει μια συνεκτική στάση σε όλη την επεξεργασία του κειμένου. Έχω κάποιες τροπολογίες εκ των οποίων ορισμένε είναι τεχνικής κυρίως φύσης. Θέλουμε εδώ πέρα να εισάγουμε λίγο περισσότερο την έννοια της συνενετικής συμφωνίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προβλεφθούν αποζημιώσεις και με διαφορετικούς τρόπους, εξοδικαστικούς. Θέλουμε λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα αυτή, να υπάρξει η δυνατότητα αυτή στο κείμενο. Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε την δυνατότητα άσκησης προσφυγής είτε από έναν είτε από περισσότερους εκπροσώπους θυμάτων παραβιάσεων της νομοθεσίας πυρενταγωνισμού. Αυτό θα πρέπει να προβλέπεται για λόγους οικονομικούς αλλά και για λόγους νομικής βεβαιότητος. Νομικής ασφάλειας μάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην καταλήγουμε σε αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις. Ξέρω ότι αυτό εναπόκειται πάλι στην διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών, αλλά ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική διάταξη και στο δικό μας κείμενο και στη δική μας την πρόταση. Επίσης, θα πρέπει να προστατεύσουμε τα προγράμματα επικούς μεταχείρισης. Πάλι θα πρέπει να πετύχουμε εδώ την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην προστασία αυτών των προγραμμάτων και τη διασφάλιση των ε, δικαιωμάτων ε, των θυμάτων, να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να ασκήσουν μια καλά τεκμηριωμένη προσφυγή. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ε, τα απαραίτητα αυτά προγράμματα ποικούς μεταχείρισης, αλλά θα πρέπει να προβλέπετε και το απαραίτητο επίπεδο ευελιξίας, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή διάκριση στις απαιτούμενες πληροφορίες για κάθε υπόθεση ξεχωριστά. καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποια τμήματα του ενημερωτικού κειμένου, των αποδεικτικών στοιχείων που μπορεί να είναι σχετικά προς μια συγκεκριμένη προσφυγή, αλλά πάλι τα οποία δεν είναι κέρια στοιχεία και τα οποία μπορούν να προστατεύονται από το απόρριτο. Τώρα, όσον αφορά τις ζημίες εκείνες που έχουν να κάνουν με μια εταιρεία αλλά και με ιδιώτες. Ξέρετε ότι θα πρέπει να υπάρχει πάλι δυνατότητα καταβολής αποζημιώση τόσο για μία ομάδα καταναλωτών όσο και προς μεμονωμένους καταναλωτές. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πρέπει να επιβάλλεται μία κύρωση δύο φορές και να αγκάζεται μία εταιρεία να καταβάλει διπλούν μία αποζημίωση. Πρέπει να, να εξασφαλίσουμε επίσης ότι δεν θα προβλέπονται κυρώσεις τιμωρητικές και ότι ε, δεν θα πρέπει να επιβάλλονται παράλληλα τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές κυρώσεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι αρχές οι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό δεν θα εξετάζουν ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία όταν ε, επεξεργάζονται τις υποθέσεις αυτές. Θα πρέπει επίσης να προβλέπεται σε κάθε περίπτωση η καλύτερη δυνατή αποζημίωση των ε, θυμάτων. Θα πρέπει όμως αυτό να γίνει αρκετά νωρίς, έτσι ώστε η αρμόδια αρχή περιανταγωνισμού να αναλάβει την κατάλληλη δράση και να μην υπάρχει καμία καθυστέρηση. Πιστεύω ότι τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην τελική εκδοχή του κειμένου. Ένα ακόμα σημείο το οποίο πρέπει να συζητήσουμε είναι οι ομαδικές κυρώσεις, οι κυρώσεις σε επίπεδο ομίλου. Νομίζω θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις συγκεκριμένες συστάσεις οι οποίες δεν θα είναι δεσμευτικές. Στην περίπτωση όμως αυτή θα καταλήξουμε τελικά σε συλλογικές προσφυγές οι οποίες θα διαφέρουν πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη. Στο στάδιο λοιπόν αυτό δεν θα πρέπει να εγκρίνουμε διατάξεις οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα πολύ διαφοροποιημένο περιβάλλον συλλογικών προσφυγών. Πιστεύω ότι όσον αφορά τη δυνατότητα συλλογικών προσφυγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρχει ένα αρμονισμένο κοινό πλαίσιο θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να επιτρέπουν την άσκηση συλλογικής προσφυγής προκειμένου να προστατευθούν τα θύματα παραβιάσεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Θα πρέπει όμως να δούμε και ποιες θα είναι οι σωρευτικές επιπτώσεις μιας τέτοιας δυνατότητας. Θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχουν κοινέ αρχές οι οποίες να ισχύουν για όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς να πρέπει να εγκριθούν συγκεκριμένοι δεσμευτικοί κανόνες αναγκαστικά για τον τρόπο διεξαγωγής και άσκησης της συλλογικής προσφυγής. Έγινε ήδη μια ανταλλαγή απόψεων, προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία και του επόμενου μήνε. Πρέπει να σα πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο από την ήδη επιτευχθήσα εργασία και από την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με την εισηγητή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ η Σόφη Ιντβελτ για του φιλελεύθερου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ τον εισηγητή, διότι όπως συνήθως συνεργάστηκε και με όλους και δεν απέκλεισε κανέναν. Όπως ε, είπε η κυρία Σάντσες Πεσέρο, υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν θα επαναλάβω. Θα ήθελα να κάνω κάποιες επιπρόσθετες παρατηρήσεις. Συχνά λέγεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια δίκαιη δίκη, δηλαδή να αποδίδεται η δικαιοσύνη στις εταιρείες που συμμετέχουν σε μια σύμπραξη, καρτέλ. Ε, και συμφωνώ, διότι έχουμε μιλήσει και για θεμελιώδη δικαιώματα επ' αυτού. Αν δούμε όμως τη διαδικασία της επίοικια, ε, τότε δεν πρόκειται για διαδικασία δίκαιη δίκαιη, διότι σημαίνει αυτό πως ένα μέρος που έχει κάνει κάτι αξιόπινο ε, έχει πλεονέκτημα ε, και λέμε στους άλλους ότι έχουν φορολογικά κίνητρα ε, οικονομικά κίνητρα μάλλον για να απορροφήσουν την τιμωρία. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι στα ε, δίκαιη δίκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτομάτως εφαρμόζει την διαδικασία επιοίκειας και θεωρεί ότι είναι μονόδρομος για τον ε, εντοπισμό των καρτέλ. Όχι, δεν συμφωνώ γιατί δεν χρησιμοποιεί άλλες ερευνητικές μεθόδους. Αυτή η διαδικασία ε, μπορεί να είναι ένα από τα μηνύματα μία μέθοδος, μία ίστατη μέθοδος ε, ε, που θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε, αλλά σίγουρα όχι μοναδική και συνιστά και παραβίαση της συνθήκης ε, κατ' εμέ το να ζητήσουμε απόλυτη απαγόρευση για τη δημοσιοποίηση. Ενώ ο γενικός κανόνας είναι η διαφάνεια. Είναι παραβίαση συνθήκης αυτό και κάποιος ε, ε, ε, είναι πάρα πολύ αποσχολημένος και μιλάει στο κινητό, Λοιπόν, δεν μπορούν να απαγορευτούν οι δημοσιοποίησεις γιατί αντιβαίνει αυτό στις συνθήκες. Οποιαδήποτε τέτοια απαγόρευση πρέπει να αιτιολογείται κατά περίπτωση. και αν το αφήσουμε αυτό στα εθνικά δικαιοδοτικά όργανα, στους εθνικούς δικαστές, Εμεί μπορούμε να δώσουμε κατευθυντήριε γραμμές, όμως κατά περίπτωση θα κρίνουν και θα αποφαίνονται οι δικαστέ σε εθνικό επίπεδο. Ο εισηγητής ε, ε, στην 158 για μια τροπολογία για το άρθρο 6 προσπάθησε να μας δώσει κάποιες τέτοιες κατευθυντήριες γραμμές. Είναι λεπτό και δύσκολο το ζήτημα. Ε, ουσιαστικά Μιλάμε για την πιθανή ανατροπή του βάρους της απόδειξης, ε, ανα, αντιστροφή του βάρους της απόδειξης Λέγεται λοιπόν ότι πρέπει κάποιο να αποδείξει ότι υπέστη μία ζημιά, αλλά πώ θα το αποδείξει άμα δεν έχει πρόσβαση στις αποδείξεις και μπορείτε να έχετε όμω λένε πρόσβαση στι αποδείξει, μόνο αν έχετε στοιχειοθετήσει ότι έχετε υποστεί ζημιά. Δηλαδή ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο τα θύματα ε, των πρακτικών επιζήμιων για τον ανταγωνισμό να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να φέρουν μια υπόθεση στα δικαστήρια γιατί ποτέ δεν θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που χρειάζονται. Χρειάζεται συζήτηση για να βρούμε λύσει για αυτά τα ζητήματα, διότι ε, ε, επί της ουσίας θα είναι αδύνατον για μικρές εταιρείε θύματα μεγάλων καρτέλ να εκινήσουν μια διαδικασία για την ε, αίτηση αποζημίωσης για ζημιά. υποστηρίζουμε, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την αρχή της συλλογική αποζημίωσης. τις συσκέψεις των σκιωδών θα δούμε εάν μπορούμε να ε, συγκλίνουμε περισσότερο για αυτό το ζήτημα. Πάντως ε, ε, το θέμα των συλλογικών αποζημιώσεων θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε διότι επιτυγχάνουμε μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην επιβολή του νόμου σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο είναι ρόλος κλειδί αυτός του κράτους στην επιβολή του νόμου, αλλά ε, ε, είναι σημαντική και επιβολή σε ιδιωτικό επίπεδο, σε επίπεδο εταιριών και ορισμένες φορές η σύγκληση είναι σχεδόν αδύνατη. Η κυρία Σάντσες Πεσέρο ε, μίλησε για ε, τα ε, πρόστιμα και τις αιτήσει αποζημίωσης. Αυτό δεν είναι αποζημίωση, είναι ε, κύρωση για κάτι το αξιόπινο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οι εταιρείε που θεωρούν ότι ε, δεν ε, τις μεταχειρίζονται σωστά, ας μην μπουν σε καρτέλ. Ε, έτσι μπορούν να αποφύγουν και τη ζημιά και άλλα δυσάρεστα πράγματα. Ας μην συμμετέχουν σε τέτοιες πρακτικές επιζήμεις για τον ανταγωνισμό. Νομίζω είναι η καλύτερη συνταγή για αυτές. Ευχαριστούμε. Για τους πράσινους. Ο κύριος Μπάσε, αλλά δεν είναι εδώ, έτσι. Ναι, ναι, εγώ παίζω τον αντικαταστάτη. Ε, ζητώ και πάλι συγγνώμη ε, εξ ονόματος του συναδέλφου που δεν μπόρεσε να έρθει. Θα ήθελα να πω ε, κάποια πράγματα στη... για αυτή την έκθεση. Ε, θετικά διακύμεθα γενικά. Ε, θα θέλαμε να κάνουμε δύο γενικόλογες παρατηρήσεις. Πρώτον, για την πλειοσφία των θυμάτων ε, τέτοιων πρακτικών επιζήμων για τον ανταγωνισμό δεν είναι δυνατό αυτή τη στιγμή συλλογικά να ασκηθεί το ατομικό ευρωπαϊκό δικαίωμα στην αποζημίωση. Ε, Επίση, σήμερα είναι σχεδόν ανέφικτο το να προσμετρηθεί το μέγεθος ε, της ζημιά επί του ανταγωνισμού λόγω των πρακτικών. Αυτό πλήττει και την εμπιστοσύνη που έχουν ε, οι πολίτες και οι καταναλωτέ στην εσωτερική αγορά. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση για ένα συναφέ ζήτημα. Εάν οι επιχειρήσεις δεν ε, αντιμετωπίσουν αυτές τις καταγγελίες των καταναλωτών μπορεί να θεωρήσουν ότι έχουν δικαίωμα να παραβιάζουν το δίκαιο ανταγωνισμού. Ο συμβασμός που εισηγείται ο εισηγητής ε, θα μπορούσε να μας βοηθήσει να υπερπηδήσουμε αυτές τις βασικές δυσκολίες. Δυστυχώς όμως οι προτινόμενες τροπολογίες δεν το επιτρέπουν στην ουσία εάν δεν προβλεφθούν μηχανισμοί ε, συλλογικών ε, δράσεων και αποζημιώσεων, collective redress ε, στα αγγλικά, δύσκολα μπορούμε να φανταστούμε με ποιο τρόπο αυτή η συμβαστική λίστα επιτρέψει, θα μας επιτρέψει να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτές τις επιζήμες για τον ανταγωνισμό πρακτικές κάποιων επιχειρήσεων. Η απουσία ε, μηχανισμών συλλογικών δράσεων για αποζημίωση de facto ευνοούν τις εταιρείες που παραβιάζουν το δίκαιο ανταγωνισμού. Εμείς ε, θεωρούμε πως ε, χρειαζόμαστε δεσμευτικές ε, δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα υπό τη μορφή συλλογικών δράσεων που διέπονται από το δημόσιο ιδιωτικό δίκαιο ε, και δεσμευτικές δράσεις επίσης από πλευράς των αρχών αρμοδίων ε, για το δίκαιο ανταγωνισμό, τόσο ώστε να αντιμετωπιστούν αυτές οι καταχρηστικές συμπεριφορές ε, και να μην υπάρχουν οικονομικά κίνητρα για την παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού. Είναι οι εισάξεις ως προς τη σημασία τους αυτές οι δύο πρακτικές και θα πρέπει να θεσμοθετηθούν στην κείμενο νομοθεσία της Ένωσης. Ο Σκιώδης που απουσιάζει θα συνεχίσει τη συνεργασία με τον εισηγητή για να εκπονηθούν εξισορροπημένες συνενετικές τροπολογίες με τρόπο ώστε να έχουμε ένα ένομο πλαίσιο που θα προστατεύει ε, τα θύματα αυτών των επιζήμιων για τον αγωνισμό πρακτικών ή δυνατόν ε, προτού εκπνεύσει η τωρινή θητεία. Okay, thank you. Um... Σας ευχαριστώ. Για τους ε, πράσινους, όχι, ε, συντηρητικούς, κυρία Πρόεδρε ναι, ναι. Σας μετακίνησα λίγο. Κυρία Πρόεδρε, θα περιοριστώ σε τέσσερα σχόλια. Μπορεί να προχωρήσει κατάπληξη σε κάποιους, αλλά είμαστε υπέρ της πρότασης της Κομισιόν. Συμφωνούμε πως πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ ε, δημόσιας και ιδιωτικής επιβολής του δικαίου του ανταγωνισμού γιατί βεβαίως ε, αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα το δίκαιο του ανταγωνισμού. Οπότε θα πρέπει να διευκολυνθεί η αποζημίωση των θυμάτων. Θα ήθελα λοιπόν να επενέσω την Κομισιόν. Η πρότασή της πρέπει να υιοθετηθεί ως έχει. Όμως είμαστε αντίθετοι με τις ε, συλλογικές αποζημιώσεις σε αυτήν εδώ την οδηγία νομίζω πως ταιριάζει καλύτερα στις συστάσεις όπως προτείνει η Κομισιόν. Υποστηρίζουμε βεβαίω τη συλλογική επανόρθωση η οποία θα πρέπει να υπάρχει στα κράτη-μέλη ε, εκεί όπου δίνει το ευρωπαϊκό δικαιο δικαιώματα σε πολίτες και εταιρείε, αλλά όχι σε αυτήν εδώ την οδηγία. Η σύσταση της ε, Κομισιόν ε, έχει στόχο να διασφαλίσει μια συνεκτική οριζόντια προσέγγιση στο ζήτημα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν προσπαθεί να εναρμονίσει τα συστήματα συλλογικών αποζημιώσεων σε ένα σύστημα το οποίο υποτίθεται θα βολεύει όλου, αλλά στην πραγματικότητα κανέναν. Θεωρώ πω κάποιε λεπτομέρειε βεβαίω χρειάζεται κάποια ρύθμιση. Έχουμε υποβάλει 10 τροπολογίε, άρα είναι σαφέ πω θέλουμε να παραμείνουμε ε, πάρα πολύ κοντά στην ε, αρχική πρόταση της Κομισιόν. Αλλά κάποιες πτυχές ε, της πρότασης έχουν εκτεταμένες ε, συνέπειες στο δικονομικό δίκαιο. Θεωρούμε πως πρέπει να διαγραφούν. Αλλά η βασική μας ανησυχία αφορά την προστασία των ε, εγγράφων επίοικιας στο πλαίσιο των ε, αποζημιώσεων στις αστικές διαδικασίες. Θεωρούμε πως πρέπει να διασφαλίσουμε πως η ιδιωτική επιβολή του νόμου δεν σημαίνει πως ε, τα προγράμματα επίοικιας θα εξασθενήσουν. Για να ανοιχνεύσουμε και να τιμωρήσουμε τα καρτέλ, οι αρχές ε, παρέχουν ασυλία ή μειωμένα πρόστιμα σε αυτούς που συνεργάζονται. Τα προγράμματα επί είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την ανείχνευση και καταπολέμηση των καρτέλ. Οι πληροφορίες που δίνουν λοιπόν οι πληροφοριδότες είναι πάρα πολύ σημαντικές, όπως και η προστασία τους. Άρα, για να διατηρηθούν τα κίνητρα συνεργασίας με τις αρχές του ανταγωνισμού πρέπει να διατηρήσουμε τις δικλείδες που προτείνει η Κομισιόν, μεταξύ των οποίων και η αποκάλυψη ε, των εγγράφων επιδικίας. Διαφωνώ με τους συναδέλφους που στόχο έχουν να εξασθενήσουν αυτές τις εγγυήσει. Έχουν κέρια σημασία για τους πληροφοριοδότες και για την επιτυχία της επιβολής του νόμου. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, αυτή στην δεν υπάρχει αναλλακτική ε, από τους πληροφοριοδότες. Τι άλλο θα κάναμε. Υποκλοπές, παρακολουθήσεις εταιριών σαν την NSA θα έπρεπε να παραβιάσουμε την ιδιωτική ζωή σε βαθμό ανεπανάληπτο. Κυρία Νετφέλτ, δεν νομίζω να θέλετε κάτι τέτοιο. Αλλά εκεί θα καταλήξουμε, εάν δεν στηρίξετε την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ. Γιούργεν, εσείς θα μιλήσετε για την ΚΟΕ, Ευχαριστώ, Σάρων. Κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, ευχαριστώ τον εισηγητή. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και την Κομισιόν. Η διαδικασία ήταν αρκετά επίπονη. Τώρα έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Οπότε οφείλουμε να ευχαριστήσουμε την Κομισιόν. Κατά την άποψή μου η πρόταση είναι εύστοχη, θα χρειαστεί, βεβαίω κάποιε τεχνικές αλλαγές, αλλά σε γενικές γραμμές είναι, όπως είπα, εύστοχη, θετική η πρόταση και πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την κατεύθυνση στην οποία πηγαίνει η Κομισιόν. Για τι συλλογικέ προσφυγέ υπόθηκαν κάποια πράγματα, επί της αρχής εγώ το θεωρώ σωστό. Το ερώτημα είναι το εάν εδώ πρέπει να ρυθμιστεί σε αυτήν εδώ την έκθεση ή, όπως είπε η Κομισιόν, να υπάρξει μια γενική οδηγία για αυτό το θέμα. Και εάν γίνει κάτι τέτοιο πραγματικά ε, σκέφτομαι πώς να το δούμε το θέμα αυτό κάπως πιο προσεκτικά ή να το αφήσουμε σε μια άλλη οδηγία. Όπως είπα, όχι γιατί είμαι εναντίον, αλλά γιατί είμαι υπέρ των γενικών ρυθμίσεων αντί του να ρυθμιστεί το ζήτημα αυτό σε πολλές μεμονωμένες οδηγίες. Γιατί μετά υπάρχει το πρόβλημα βεβαίως ε, αντιφατικών διατάξεων. Για τους λόγους που ανέφερα. Στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν. Δεν ε, έχουμε υποβάλει άρα τροπολογίες, αλλά θα θέλαμε να δούμε την ε, όλη εξέλιξη του θέματος και αναμένουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Μίλησαν οι σκιώδες συγητές. Κάποιος άλλος. Ναι, Hans Peter Martin. Ναι, ναι. Κάπου εδώ ήτανε. Μου διέφυγε. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, με έχουν καλύψει προαλήσαντες. Δύο γενικές παρατηρήσεις. Αφού μιλάνε περισσότεροι γερμανικά, ας μιλήσω και εγώ γερμανικά. Είναι ένα νομοθετικό μέτρο το οποίο είναι πάρα πολύ γενικά και ευρύτατα διατυπωμένο. Θεωρώ πως ε, στα ζητήματα αυτά θα πρέπει να εργαστούμε περισσότερο στο μέτωπο του Λακωνίζιν. Επίσης είδαμε πως ε, έχουμε διάφορα ε, σχόλια που προέρχονται από διάφορα συμφέροντα. Για το θέμα λοιπόν του νομοθετικού αποτυπώματος, καλό είναι να ξέρουμε από πού προέρχονται αυτές οι προτάσεις. Δηλαδή, πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν καλές ιδέες, αλλά θα πρέπει να τα ξέρουν αυτά και οι ψηφοφόροι. Okay, uh, as I managed to put Μια που κατάφερα να υποβάλω 46 τροπολογίες, σας πω και εγώ κάτι. Ουσιαστικά στις ε, τροπολογίες μου ακολουθώ τα όσα είχαμε πει στην Επιτροπή μας στο παρελθόν. Δεν θα σας ε, προξενήσουν καμία έκπληξη. Να τονίσω απλώς κάποια στοιχεία για ένα συγκεκριμένο σημείο όσον αφορά τα εις δημόσιες κυρώσεις για τη μετακύληση των επιπλέον επιβαρύνσεων. Ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλω εδώ να διασφαλίσω είναι ότι οι κυρώσεις αυτές μπορούν να θέσουν εκτός αγοράς μια επιχείρηση και προφανώς αυτό δεν πρέπει να γίνει για την προστασία αν μη τι άλλο των θέσεων απασχόληση. Ωστόσο συμβαίνει ορισμένες φορές αυτό το πράγμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν λαμβάνει κανείς καμία απόλυτο αποζημίωση. Ήθελα απλώς να τονίσω το ζήτημα αυτό να φωτίσω την πτυχή αυτή και νομίζω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα καταβολής της αποζημίωσης σε ένα μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε η καταβολή της αποζημίωσης να λειτουργήσει τελικά κατά της ίδιας της εταιρείας και των καταναλωτών. Όσον αφορά τώρα την προστασία των δεδομένων στα πλαίσια των προγραμμάτων επικούς μεταχείρισης, η ισορροπία εδώ είναι πολύ λεπτή νομίζω θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και εμείς στη διατύπωσή, στη μας. Σε ορισμένε περιπτώσεις όντως θα πρέπει να κοινοποιηθούν, να οι πληροφορίες αυτές. Διαφορετικά οι καταναλωτές ε, μένουν εκτεθειμένοι και δεν μπορούν να λάβουν την ε, κατάλληλη αποζημίωση. Και πάλι όμως νομίζω ότι μπορούν να υπάρχουν εδώ πέρα πολλές διαφορετικές αποχρώσεις και αυτές ακριβώς προσπαθώ να τονίσω με τις τροπολογίες μου. Τώρα, όσον αφορά τις προθεσμίες παραγραφής. Νομίζω ότι πρέπει να προβλεφθεί ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εδώ πέρα α, χρησιμοποιώ την χρονική περίοδο που προβλέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αν θέλετε είναι η χώρα με τις περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις, προσφυγές δηλαδή για ζητήματα ανταγωνισμού. Νομίζω λοιπόν ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια χρονική περίοδο, άλλωστε έχουμε δοκιμάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο αυτή, λειτουργεί καλά, το ότι προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαστικά κακό. Η μετακύληση των επιπλέον επιβαρύνσεων είναι νόμιμη, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ενδεχομένω η μετακύληση της αποζημίωσης στην αλυσίδα εφοδιασμού μπορεί να αποβεί αρνητική και επιζήμια τελικά, οπότε εγώ προσπάθησα να βελτιώσω εδώ κάπως την κατάσταση. Δεν θέλω να μετακινήσω την, το βάρος της απόδειξης, αλλά νομίζω ότι οι προτάσεις που κάνω από εμπορική πλευρά είναι λογικές. Νομίζω λοιπόν ότι η πρόταση που γίνεται είναι θετική για τη μετακύληση αυτή από τη μία εταιρεία στην άλλη, από τον έναν καταναλωτή στον άλλον. Άλλωστε η ε, εταιρεία η οποία συμμετέχει στην ακαρτέλ γνωρίζει τελικά αν έχει συμβεί ή όχι μια εταιρεια στην αλλη απο τον εναν στον αλλον αλλωστε η εταιρεια η οποια μετακύληση. Σας προτείνω επίσης να έχουμε έναν υποχρεωτικό μηχανισμό συνενετικής ε, διευθέτησης, ο οποίος ε, δεν θα είναι αναγκαστικά δεσμευτικό αν το αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, αλλά καθότι προωθούμε γενικότερα τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης και διευθέτησης, είναι σημαντικό και εν προκειμένου να προβλέπετε μια τέτοια δυνατότητα. Και στις τροπολογίες μου έχω υποβάλει κάποιες παρατηρήσεις που συνάδουν με τόσο είπαν οι προλύσαντες. Προσπαθώ πάντως να βρω κάπως την ε, μέση οδό ανάμεσα σε αυτό το οποίο εγώ πραγματικά θα ήθελα, δηλαδή πιο ισχυρή στάση σε ορισμένα σημεία και ανάμεσα στην αναζήτηση μιας συμβαστικής λύσης για άλλα σημεία. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο, αν όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Δεν νομίζω Ναι, μπορείτε να πάρετε το λόγο σύντομα όμως παρακαλώ. Ευχαριστώ και θα είμαι σύντομο. Όπω είπε και ο κύριο Φαμπ, επιβεβαιώνω ότι κατά την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν συντρέχει λόγο να τροποποιηθεί η νομική βάση ε, και με χαρά θα συνεχίσουμε τη συνεργασία για αυτό το νομοθέτημα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διάσκεψη των Πρόεδρων ανέλαβε δέσμευση προ μεγάλη μα ε, ικανοποίηση να περατώσει τη διαδικασία προτού διεξαχθούν οι επόμενε ευρωπαϊκέ εκλογέ και με τα χαρά θα δεχτούμε με την πρόσκληση του κυρίου Σφάμπ να συζητήσουμε όλοι μαζί με τον εισηγητή και του κοιόδης ε, τι διάφορε πτυχέ ε, τη νομοθετική πρόταση, γιατί από ό,τι κατάλαβα διάφοροι ευρωβουλευτέ ανησυχούν για το ρόλο, τον ενδεχόμενο ρόλο της αρχής επίοικιας για τη δημόσια επιβολή του νόμου και πώ μπορούμε να επιτύχουμε την βέλτιστη ισορροπία με την επιβολή του ε, δημόσιου ιδιωτικού δικαίου. Αντρέα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε και η συνάδελφος. Προσκαλέσαμε την Κομισιόν. Κύριε Μάρτιν, κάναμε μια ακρόαση όπου ακούστηκε, ακούστηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ήταν πολύ διαφανής η διαδικασία και στο πλαίσιο των εκθέσεων που κάνουμε για τον ανταγωνισμό Ήμουν και εγώ εισηγητής, ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο ήταν εισηγητής, ο κύριος Τρεμόζα είχε ασχοληθεί με αυτή την έκθεση. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά στοιχεία που είχε οθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε ήταν διαφανής η διαδικασία. Αλλά θα ήθελα να πω πως υπάρχουν αφενός γενικά επιχειρήματα, όπως παραδείγματος χάρη να ε, συμφωνήσω με τον κύριο Μάρτιν στο να μην είναι τόσο δυσνόητο το κείμενο, αλλά βεβαίως ε, οι λεπτομέρειες έχουν μεγάλη σημασία. Τώρα για αυτό το οποίο είπε η κυρία Ινετφέλντ, πως ε, δεν υπάρχει η αρχή της δικής δίκης. Πρέπει να πούμε πως νομικά εδώ πέρα δεν είναι ποινική η διαδικασία, οπότε πρέπει να ισχύουν οι ίδιες αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται παντού. Ε, μα ούτως ή άλλως ε, και στο ποινικό δίκαιο ακόμα η μεταμέλεια αποτελεί παράγοντα επίοικιας, οπότε δεν ε, είναι τόσο φοβερά τα πράγματα. Αλλά η ποινή μπορεί να μειωθεί και σε αυτή την ε, περίπτωση νομίζω. Δεύτερον, βεβαίω έχουμε κάποια θέματα στα οποία συμφωνούμε με την Κομισιόν. Χαίρομαι πως είπε ο κύριος Κλούτε πως ε, ε, πρόκειται για τεχνικές μικρορυθμίσεις και ο κύριος Έπινγκ τώρα έχει κάνει 10 τροπολογίες. Αν είναι αυτές οι μικρορυθμίσεις που θέλουμε δεν το ξέρω, αλλά το ECR πράγματι έχει κάνει κάποιες ενδιαφέρουσες ε, τροπολογίες που μπορούσαν να βελτιώσουν τα πράγματα. Τώρα η Κομισιόν εδώ πέρα αφενός έχει τα στοιχεία της ε, συλλογική ε, προσφυγής σε μια σύσταση προς το Συμβούλιο και από την άλλη βεβαίως έχουμε τα άμεσα ζητήματα που μπαίνουν σε μια οδηγία και είναι νομίζω σωστό αυτό. Γιατί, γιατί κυρία Πρόεδρε βρέπουμε κάποιες διαφορές ε, μεταξύ των ε, κρατών μελών που προσπαθούν, όπως είπα, ε, για λόγους και οικονομίας χρόνου και στα δικαστήρια να ομαδοποιήσουν συχνά τους ενάγοντες αλλά όπως είχαμε δει και πριν από λίγα χρόνια στη Γερμανία σε μια περίπτωση πάρα πολλών αναγώνων κατά της ε, Deutsche Telekom δεν είναι τόσο απλό κάτι τέτοιο οπότε προσπαθούμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα για να έχουμε και διασυνοριακές τέτοιες ε, προσφυγές γι' αυτό θεωρώ πως ε, πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου πως πάντα η Κομισιόν έκανε το διαχωρισμό αφενός ε, συλλογικές πρόσφυγες ε, στο επίπεδο των κρατών και από την άλλη ευρωπαϊκό, κάποια ευρωπαϊκή εναρμόνιση στο επίπεδο του δικαίου. Το ένα είναι αυτό. Το ζήτημα τώρα του τι κάνουμε με τα έγγραφα που δίνουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες και, αν και βεβαίως βοηθάνε έτσι άμεσα τους καταναλωτές και τις άλλες επιχειρήσεις. Με αυτά τα οποία λέει η Κομισιόν, μπορεί να ξεκινήσει όλη η διαδικασία εάν ξεκαθαρίσει νομικά και διοικητικά πως τα έγγραφα αυτά τελικά είναι προστατευμένα. Και έτσι μετά η Κομισιόν παρέχει πρόσβαση στα σημεία εκείνα τα οποία είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Βεβαίω η Κομισιόν στο άρθρο 6 παράγραφος 1α και β τι κάνει. Παρέχει μία απόλυτη προστασία στα έγγραφα τα οποία θα χρησιμοποιήσει η ίδια. Η, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις δύο υποθέσεις που ε, προανέφερα έκρινε το θέμα αυτό και είπε πως δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Στην Πρίζ λοιπόν είχαμε μια διάσκεψη σχετικά και ένας δικαστής του ΔΕΚ είπε πως τελικά υπάρχει η δυνατότητα αυτής της ε, προστασίας, ε, θα μπορούσε να υπάρχει στον νόμο. Οπότε εγώ κατέληξα στο ότι ένας δικαστής πρέπει να αξιολογήσει την υπόθεση και μετά ένα-ένα τα έγγραφα. Αφενός ως προς το συμφέρον ε, των ε, εναγόντων και βεβαίω ε, και από τη σκοπιά του προστατευόμενου μάρτυρα για να κρίνει το εάν θα προστατεύονται τα έγγραφα ή όχι. Τώρα δεν ξέρω εάν οι τροπολογίες οι οποίες μοίρασα και στον κύριο Μπάς Αϊκχάουτ ε, σας ικανοποιούν δεν είναι συμβαστικές, είναι η δική μου η άποψη ούτως ή άλλως. Ε, ήδη για το άρθρο 6 έχω στείλει μια πρόταση συμβιβαστική όπου προσπαθώ να δώσω μια καθοδήγηση, αν θέλετε, στην ε, διαδικασία αξιολόγησης των εγγράφων και ε, να υπάρχει η δυνατότητα να κρίνουμε το κάθε έγγραφο μονομένα πόσο σημαντικό είναι για την προστασία της, ε, του μάρτυρα, για την αποκάλυψη του καρτέλ και βεβαίως η οδηγία αυτή ε, καθορίζει μόνο την διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Αυτή είναι η σημασία γιατί η κυρία Ινετφέλντ είπε πως έχει μετά ο μάρτυρα συμφέρον ε, να φέρει τους φακέλους για να θεμελιώσει αυτά τα οποία λέει πράγματι, αλλά αυτά πρέπει να τα πάει στην Κομισιό, να υπάρχει μια γενική εικόνα, ενώ εδώ πέρα μιλάμε για την πρόσβαση στα έγγραφα, στην αστική διαδικασία, μετά την ε, εκδίκαση της ε, ποινική ε, υπόθεσης. Οπότε αν δημιουργήσουμε όπως είπα νέους κανόνες θα πρέπει να καλύπτουν και το τι γίνεται με τη διαχείρισή τους από την και το τι γίνεται στην δίκη. Μετά για το ζήτημα της περαιτέρω διάδοσης ε, των εγγράφων αυτών. Κοιτάξτε, εάν υπάρχει όπως σας είπα αυτό το οποίο λέει ο καθηγητής ε, Μπονκαμ του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου για την μετακύληση των ε, επιβαρύνσεων στην περίπτωση στην οποία κάποιοι προσφεύγουν σε δικαστήρια σε διαφορετικές χώρες, ε, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα υποχρεωτικά να πάνε όλες αυτές οι υποθέσεις να εκδικαστούν μαζί σε ένα σημείο. Και θα μπορούσαν να ε, να είναι επιτυχής οι δίκες γιατί δεν μπορεί κάποιος να αποδείξει πως ε, ε, ο ενάγων ε, είχε, δεν είχε δυνατότητα να μετακυλήσει την επιβάρυνση. Εδώ πέρα λοιπόν ο συνάδελφος ο κ. Σάντσες Πρέσεδο έχει κάνει μια αρκετά ενδιαφέρουσα παρέμβαση, αλλά οπωσδήποτε συμφωνούμε πως θα πρέπει να μειώνεται η επικάλυψη της επιβάρυνσης. Οπότε αυτό το οποίο προτείνει ο κύριος Σαντσπρεσέζο αυτή τη στιγμή δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες γιατί το εάν έχει υπάρξει κάποια μετακύληση ή όχι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρουν όλοι οι δικαστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν το εάν θεμελιώνει αυτό το οποίο λέει ο Ενάγων. Ανεξάρτητος τι μπορεί πιθανώς να αποφασιστεί σε άλλα δικαστήρια. Δεν θα ήθελα τώρα να πω άλλα να μακρηγορήσω περτέρω. Υπάρχει το ζήτημα της κοινή και αλληλεγγύας ευθύνης, υπάρχει το ζήτημα των προθεσμιών που προτείνει η Κομισιόν, ζητήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε, αλλά νομίζω κυρία Πρόεδρε πως τα επιχειρήματα των συναδέλφων έχουν ληφθεί υπόψη και αυτό το οποίο προτείνει ο κύριο Σάντσης εδώ οπωσδήποτε θα μα οδηγήσει σε κάποια λύση, αλλά η λύση αυτή πρέπει να είναι λογική και να είναι προ το συμφέρον και των καταναλωτών, αλλά και του συστήματο για να μπορεί να ανακαλύπτει τα καρτέλ των συντομότερο δυνατόν και η ισορροπία την οποία ανέφερα νομίζω είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. και για να έχει τη ναι. δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακαλύπτει καρτέλ και με τη χρήση αυτής της επίοικες όπως είπαμε. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Στις 5 Δεκεμβρίου σκοπεύουμε να ψηφίσουμε, έτσι δεν είναι. Θα χρειαστεί να αναβάλουμε όμως την ψηφοφορία μέχρι πότε. Α, είναι σαν ανακοινώσει που δεν διάβασε, αφού δεν ε, υπήρχαν εδώ αρκετοί για να με ακούσουν. Πρέπει τώρα να πάω στι ανακοινώσει μου. No, we haven't got a proposed new date, but... Δεν έχουμε προτινόμενη ημερομηνία, τέλος πάντων. Θα σας το μοιράσουμε, θα το στείλουμε. Προφανώς, στο μέτρο που θα είναι έτοιμη η η γνωμοδότησή μας προς την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, μπορεί να χρειαστούμε και περισσότερο χρόνο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα στις 27 Ιανουαρίου προβλέπεται. Η νέα πιθανή ημερομηνία είναι 27 Ιανουαρίου, λοιπόν, μέχρι νεοτέρας. Ε, για να περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης, ε, ασφάλιση έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, Σάμπο Τέρχο, εισηγητής, ε, τον είδα πριν από λίγα λεπτά, που είναι Σάμπο. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες. Εν γέννη ήταν επικοδομητικές τροπολογίες και αποσκοπούν στη βελτίωση της έκθεσης. Δεν χρειάζεται πλέον σε αυτό το στάδιο να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα παρόλα αυτά εντάχει να αναφερθώ στις βασικές αρχές. Ήδη από την πρώτη συζήτηση συνειδητοποίησα ότι υπάρχει κοινή αντιλήψη ότι δεν χρειάζεται ισχυρή εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η ανταλλαγή βελτίωση των πρακτικών μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. επίση. Ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να αποφευθεί μεγαλύτερος κίνδυνος μέσω αυτής της ανταλλαγής και οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές καλύπτονται από δύο διαφορετικά είδη ε, ασφαλίσεων που δεν πρέπει να συγχέονται δεν πρέπει να συγχαίουμε μάλλον. Για τις ε, τροπολογίες έχουμε αυτές που ασχολούνται με την αρχή της πρόληψης, τη αρχή ασφάλειας, την ενημέρωση, καθώς και με την προσθήκη παραδείγματων, όπως οι 15 και 63. Αντιτάσσομαι σε κάποιες τροπολογίες, γιατί ε, δεν θεωρώ ότι είναι ε, σκόπιμο να επαναλαμβάνουμε κάποιες αρχές που έχω ήδη συμπεριλάβει στην έκθεσή μου. Επίσης, ε, στη προκειμένη περίπτωση ε, δεν μπορώ να υποστηρίξω τις τροπολογίες που είναι υπέρ της εναρμόνισης γιατί ε, δεν ε, ισχύει δεν υπάρχει μία μαγική λύση για όλα τα ζητήματα και υπάρχουν και κάποια άλλα μεταφραστικά ζητήματα, οπότε θα ήθελα διευκρίνηση για τις ακόλουθες τροπολογίες. Τροπολογία 1 του κυρίου Λάγκε, 2 Βίσεψ και 4 Τούρβαλτς. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το περιεχόμενο των τροπολογιών. Ήδη έχω προετοιμάσει συμβαστικέ τροπολογίες και τι έχω στείλει στους Ε, Και περιμένω με ανεπομονησία να ακούσω τις απόψει και τα σχόλιά σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Βέρνερ Λάγκερ, λοιπόν, για το ΕΛΚ. Ε, ευχαριστώ τον Σίτη. Θεωρώ πως 68 τροπολογίες δείχνουν πως η έκθεση είναι καλή πως θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες, κάποιες σημεία συμφωνίας, αλλά τις συμβαστικές προτάσεις που λέτε δεν τις έχω δει ποτέ. Πότε προβλέπονται. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Δεν είναι δραματική η κατάσταση. Το ότι δεν τη είδα εγώ δηλαδή, εντάξει. Έχουμε χρόνο. Θεωρώ πως ο στόχος Κομισιόν είναι σωστός. να αυξηθεί η διάδοση των ασφαλιών ακινήτων από τέτοιες ε, καταστροφές. Είχαμε πολλές πλημμύρες τα τελευταία χρόνια. Εδώ πέρα βεβαίως ε, οι ενδιαφερόμενοι είναι ιδιοκτήτες, ε, ασφαλιστικές εταιρείες και φορολογούμενοι και βεβαίως η αξιολόγηση κινδύνου είναι ένα θετικό όσον αφορά την άμυνα απέναντι σε καταστροφές. Τώρα το να είναι τυποποιημένα τα ασφάλιστρα δεν ξέρω αν έχει νόημα. Κατόπιν. Το τι γίνεται με τις ασφαλιστικές εταιρείε που είναι offshore και τρίτον βεβαίως ε, η πρόταση της Κομισιόν για κρατική ε, για το ότι η κρατική αποζημίωση σε πληγέντες είναι ένα είδος επιδότησης και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται. Έχω υποβάλει τροπολογίες εδώ πέρα και τέρτον. Πως ε, μία αυτόματη και υποχρεωτική ασφάλιση βεβαίως αποκλίνει από τις αρχές ατομικής ευθύνης και θα είναι και πάρα πολύ ακριβή και άρα θεωρώ πως με βάση τις 66 ε, τροπολογίες ε, μπορούμε να βρούμε μια κοινή γραμμή και να επιτύχουμε καλύτερη προστασία για τους πολίτες. Να θα απλοποιηθούν οι ασφαλιστικές συμβάσεις. Ο κ. Σίγητης λοιπόν έχει υποβάλει μια καλή έκθεση και ε, ελπίζω και με τη στήριξη του ΕΛΚΑ να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ωραία. Για τους σοσιαλδημοκράτες, Άντολιν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες σύντομες παρατηρήσεις Εξ ονόματος κυρίας Μίτση, η οποία δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα το απόγευμα, ουσιαστικά θέλει εξ ονόματός της να πω το ακόλουθο. Ευχαριστεί καταρχάς τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους που έχουν συμβάλει για την βελτίωση της έκθεσης αυτής. Οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, που υποβλήθησαν σήμερα στην έκθεση αυτή αποτελούν μια καλή συνέχεια της συζήτησης που κάναμε στα πλαίσια της Επιτροπής μας στο παρελθόν και κατά την άποψή της δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα ως προς την έβρεση συμφωνίας και συμβαστικών τροπολογιών. Πιστεύει ότι οι τροπολογίες οι οποίες ε, ζητούν ε, μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική όσον αφορά ε, την ασφάλιση για τις φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές είναι σημαντικέ τροπολογίε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ενημέρωση, όσον αφορά το βαθμό διείσδυση, όσον αφορά τα ασφάλιστρα τα οποία χρεώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείε προς τους καταναλωτές. Ξέρετε ότι οι σχετικές πληροφορίε αποκλείουν πάρα πολύ από τη μία χώρα στην άλλη, επομένω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Ορισμένες τροπολογίες επίσης αναφέρονται στην ιδέα της ατομικής ευθύνης. Η κυρία Μίτση θεωρεί ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τη δική τους εθνική πολιτική πρόληψη των καταστροφών, δεν προωθούνται αρκετές τέτοιες προληπτικές πολιτικές και πολύ συχνά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλήρης εφαρμογή των σχετικών νομικών διατάξεων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επιτελείται πολύ μεγαλύτερη ζημιά κατά αυτόν τον τρόπο. Επομένως, η κυρία Μίτση θέλει να υποστηρίξει τον, ιδιαίτερα την πτυχή της πρόληψης, τις πολιτικές που θα πρέπει να προωθηθούν και θεωρεί επίσης ότι δεν θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση και συμβαστικές τροπολογίες, επομένως βλέπει σε μια θετική κατάληξη για την έκθεση αυτήν. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίλς, εξ ονόματος των Φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πολιτική μου ομάδα δεν έχει να κάνει πάρα πολλές παρατηρήσεις. Θεωρούμε ότι το σχέδιο έκθεσης είναι πολύ καλά ισορροπημένο και έχω υποβάλει δύο μοντροπολογίε καθότι δεν έχουμε πάρα πολλές ανησυχίες. Για ποιο λόγο ασχολούμεθα εδώ πέρα με τις φυσικές καταστροφές και τις ανθρωπογενείς καταστροφές στο ίδιο κείμενο. Ενδεχομένως να πρέπει να προβλεφθεί και μία τρίτη κατηγορία, νομίζω την έφερε ήδη την προηγούμενη φορά, θα μπορούσε να είχαμε μία οδηγία για τις καταστροφές που προκαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά αυτόν τον τρόπο θα είχαμε μια πιο σφαιρική εικόνα της κατάστασης. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένα τις φυσικές καταστροφές. Σε αυτό αναφέρθηκε ο κύριος Τέρο. Στις φυσικές καταστροφές δεν υπάρχει η έννοια του υπευθύνου, του αυτού που φέρει δηλαδή την ευθύνη. Έτσι λοιπόν σε μια σχετική τροπολογία λέω ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου την εργασία των υπόλοιπων γενικών διευθύνσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να γνωρίσουμε επίσης ε, τι κάνουν οι υπόλοιπε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Νομίζω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή μια οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη και νομίζω και για την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση τη πυρηνική ενέργεια. Οι πρωτοβουλίε αυτέ νομίζω ότι ε, σχετίζονται και με τη δική μας την έκθεση Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει εμεί με τη δική μα την έκθεση να επαναλαμβάνουμε πράγματα τα οποία ήδη λέγονται ή ήδη ισχύουν σε άλλε εκθέσει ή άλλε οδηγίε. Πέρα από αυτά, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα με τη βοήθεια του εισηγητή του κυρίου Τέρο. Δεν έχω καμία ανησυχία. Εκτό βέβαια και από τα όσα πρέπει να δούμε στα πλαίσια των των καταστροφών προκαλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε, ε, προσωπικές παρατηρήσεις θα ήθελα να καταθέσω σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Τέρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς για τις ε, συμβαστικές του προτάσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν εν γέννη αποδεκτές, αλλά κατά την άποψή μας ε, δεν είναι επαρκής. Νομίζω ότι υπάρχει μια σημαντική έλλειψη συμφωνίας ανάμεσά μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα που μας διαχωρίζουν. Θεωρώ ότι οι τροπολογίες του δεν είναι αρκετά φιλοευρωπαϊκές, δεν περιέχουν μια σημαντική ευρωπαϊκή φιλοδοξία, δεν θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε μια εναρμόνιση ευρωπαϊκή όσον αφορά την ασφάλιση έναντι καταστροφών. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει ακριβώς προς αυτό να στοχεύουμε, μεγαλύτερη σύγκληση δηλαδή όσον αφορά την προστασία εναντί αυτών των κινδύνων, εναντί αυτών των καταστροφών που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Προτείνουμε λοιπόν κάποιες σχετικές τροπολογίες και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα εξής στοιχεία. Ο βαθμός διείσδυσης θα πρέπει να συμπληρώνεται από έναν δείκτη συμμόρφωσης των προγραμμάτων ασφάλισης σε σχέση με τους κινδύνους. Οι κίνδυνοι, οι ανθρωπογενείς είναι πολλές φορές διασυνοριακοί. Αυτό είδαμε άλλωστε και πρόσφατα στις πλημμύρες στο Δούναβι. Επομένως, η δική μας αντίδραση θα πρέπει να είναι ακριβώς διασυνοριακή, όπως και κίνδυνη. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο χρειάζεται μια ευρωπαϊκή εναρμόνιση όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνονται προς τους ασφαλισμένους προτού συνάψουν μια τέτοια συμφωνία ασφάλισης. Πρέπει επίσης να έχουμε μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων όσον αφορά τις επικίνδυνες γεωγραφικές ζώνες και να έχουμε για τις βάσεις αυτές δεδομένων διαδραστικά διαδραστικές ιστοσελίδες. Χρειαζόμαστε επίσης ανάληψη περαιτέρω δράσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις εθνικές αρχές για να δίνονται περισσότερες πληροφορίε προς τους καταναλωτές. Μου ζητήσατε κύριε Τέρο περαιτέρω εξηγήσει για την τροπολογία παριθμών 12, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν την καταλαβαίνετε πολύ καλά. Η τροπολογία αυτή δεν πρόκειται να διαβάσω αυτή τη στιγμή. Τι λέει ουσιαστικά, ότι ε, η, τα σύνορα μεταξύ φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα δύο αυτά είδη καταστροφών είναι όλο και πιο ασαφής. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι οι φυσικές καταστροφές οξύνουν και διευρύνουν τις ζημίες των ανθρωπογενών καταστροφών. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο οφείλουμε να προσεγγίζουμε τα πράγματα πιο σφαιρικά. Αυτό λέει η τροπολογία. Σας ευχαριστώ. Thank e Σας ευχαριστώ, Άσλε, για τους συντηρητικούς. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Η αρχική έκθεση ήταν πολύ καλά διατυπωμένη. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπεζέ, εγώ δεν θεωρώ πως χρειαζόμαστε ισχυρή ευρωπαϊκή παρουσία στον τομέα αυτών. Υποστηρίζω τις περισσότερες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί, οι περισσότερες από αυτές είναι πολύ ισορροπημένες και θεωρώ πως ε, εθνικές, με φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές ε, είναι κάτι που πρέπει να δούμε χωριστά και διαφέρει και η αντίδραση ανάλογα με την κάθε περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές τροπολογίες ζητάνε προληπτικά μέτρα σε επίπεδο κράτους, μέλους ε, και περιφέρειας, με το οποίο, κάτι με το οποίο συμφωνώ, γιατί τα κράτη-μέλη νομίζω παίζουν ένα ρόλο κλειδί εδώ πέρα και στην ενθάρρυνση της υπεύθυνη συμπεριφοράς. Είναι θετικές αυτές οι τροπολογίες καθώς αναγνωρίζουν πως δεν υπάρχει μία ενιαία λύση. Οφείλω να πω πω ανησύχησα λίγο για τη διατύπωση μια τροπολογία που μίλησε για τοξικά ασφαλιστικά προϊόντα. Λίγο προσβλητικό αυτό και ελπίζω ο εισηγητής να μην το συμπεριλάβει. Αλλά κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως η αρχαίοι ήταν αρκετά καλή. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τις περισσότερες τροπολογίες και θα βελτιωθεί έτσι το αρχικό κείμενο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ δεν βλέπω κάποιον από την Γκουέ. Ο Βέρνερ θέλει να πει κάτι. Ναι, ξέχασα κάτι. Η τροπολογία 1. Εκεί στα αγγλικά το είδαν εδώ πέρα οι συνεργάτες μου και το επαλήθευσα και εγώ, έχω πει στα γερμανικά ανάγκη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, πιθανώς ε, το, το οποίο έχει μεταφραστεί στα γερμανικά ιδιαίτερα ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο κάπως ε, διαφέρει με από το αρχικό μου κείμενο αυτό. Να μην πω ότι είναι και το αντίθετο. Αν μπορείτε να το αλλάξετε σας παρακαλώ. Αυτά για την διατύπωση. Μάλιστα, κατάλαβα. Δηλαδή κάτι πιθανώς αντί για ιδιαίτερα έπρεπε να πούμε. Ήταν κάτι το δυνητικό. Μάλιστα. Ο Σάμπο θα το σημειώσει. Ωραία, η τροπολογία σας. Η τροπολογία 1. Η δική σας τροπολογία 1. Η πρώτη τροπολογία του κύριου Λάγκεν, μάλιστα. Κάποιος άλλος. Ωραία, οπότε Σέμπο έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κυρίως για τις διευκρινήσεις. Ε, προσβλέπουμε ανυπομονησία στην επόμενη συνεδρίαση των ε, σκιωδών. Ελπίζω να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Ο στόχος μου ανέκαθεν ήταν να έχουμε ένα σύντομο κείμενο όπου ε, ξεκάθαρα φαίνεται ποια είναι η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δίνουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στην πράσινη βίβλο της Επιτροπής. Είμαι αισιόδοξο πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που να πληρεί αυτές τις προδιαγραφές. Πρόεδρος, ευχαριστώ και χαίρομαι που όλα βαίνουν αισίως. Στην Επιτροπή σκοπεύουμε στις 17 Δεκεμβρίου να ψηφίσουμε. Ε, φαίνεται ότι θα είναι δυνατό αυτό, όπως εξελίσσουν τα πράγματα και στην πρώτη ολομέλεια του Φεβρουαρίου θα ε, εξεταστεί στο Στρασβούργο. Αυτά για σήμερα. Αύριο το πρωί ανταλλαγή απόψε με τον Άγγελ Γκορία, Γενικό Γραμματέα του ΩΣΑ. Και μπορώ να σας πω ήδη από τώρα ότι συνήθως αξίζει τον κόπο. Ελπίζω να είσαστε όλοι εδώ και να περάσουμε όλοι ωραία. Τα λέμε εσάδια.